Καλημέρα, σας ε, καλωσορίζω όλους ε, στην τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές ε, διακοπές. Έχετε μπροστά σας την ημερήσια διάταξη. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παρά να την εγκρίνετε. Αυτό είναι το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης. το σημείο 2 Πάμε στην έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Ε, έχετε μπροστά σας τα πρακτικά και αν μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης ε, δεν έχετε εκφράσει την αντίρρησή σας, εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός τσεχικά, ε, λιθουανικά, μαλτέζικα και σουηδικά. Ε, νομίζω όλες οι άλλες γλώσσες, ε, για όλες τις άλλες γλώσσες προσφέρεται διερμηνία, ταυτόχρονη διερμηνία. Χαίρομαι που έχουμε εδώ τον κύριο Ντένις Κόλλη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ε, της διοργανικής επιτροπής για την παιδεία και τον πολιτισμό. Είναι ο διάδοχος του κύριου Σόιμπελ, τον οποίο την τελευταία φορά αποχαιρετήσαμε ήταν ε, πολύ σημαντική η δική του η παρουσία για τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεργασία θα είναι πολύ δύσκολη κατά τους επόμενους μήνες, γι' αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Εμείς όμως είμαστε πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι και αν είσαστε και εσείς συμπαθητικοί φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε πολλά προβλήματα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, κύριε Γκρόουλη, σας καλωσορίζουμε. Είστε Βρετανός, Ιρλανδός, τι είστε. Α, Ιρλανδός. Πολύ ωραία. Πάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ υπουργού και αναπληρωτή υπουργό, ε, γιατί ο υπουργό είναι άρρωστο, έχουμε την κυρία Καταρτσίνα Χολ. Είναι υπουργό ε, Εθνικής Παιδεία. Την κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα είναι υπουργό Επιστημών και Ανώτερη Εκπαίδευση. Τον κύριο Μπόκταν Σντρογκεύσκη, Υπουργό Πολιτισμού και Εθνική Εκκληνομιάς Νομίζω όμω δεν είναι ο ίδιο εδώ. Ε, έχουμε τον αναπληρωτή του και έχουμε τον κύριο Άταμ Κίρς, Υπουργός Αθλητισμού και Τουρισμού. Λυπάμαι που εκτός από τα μέλη του ΕΛΚ, τα οποία είναι το οποίο ΕΛΚ εκπροσωπείται ικανοποιητικά και εκτός από τον συνάδελφό μου από την αριστερά ε, δεν έχουμε άλλους ευρωβουλευτές από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και θα ήθελα τους συνεργάτες τους να τους υπενθυμίσουν ότι σήμερα έχουμε συνεδρίαση. Φαντάζομαι ότι τα μέσα στην Πολωνία θα έχουν ανακοινώσει ότι ο Πρωθυπουργό σας, ε, η παρουσία του Πρωθυπουργού σας ε, στην Ολομέλειά μας ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη. Τον ε, δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Η ομιλία του διαπνέεται από ιδιαίτερο φιλευρωπαϊσμό και θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι συνεργάτες του, ε, τους οποίους ε, μας στέλνει και συνεδριάσει μας, ε, διακατέχονται από τον ίδιο άκρατο φιλοευρωπαϊσμό. Έχουμε τον συνάδελφο Πίσες Αξέλα κοντά μας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του για την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό. Έχουμε την κυρία Χάνιμπαλ, η οποία δυστυχώς δεν είναι ακόμα εδώ, η οποία όμως θα παρουσιάσει την έκθεσή της για την κατάσταση σχετικά με ε, τους ε, μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Έχουμε τον κύριο Μπόρις, ο οποίος ε, θα παρουσιάσει τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στη ψηφιακή εποχή, την οποία έκθεση θα ψηφίσουμε τον Οκτώβρη. Και γι' αυτό έχουμε και σήμερα την ακρόαση. Έχουμε και την κυρία Παλιαδέλη, που δυστυχώς και αυτή δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι η συγγήτρια για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Όπως ξέρετε, η έκθεση αυτή, το θέμα αυτό ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της Ουγγρικής Προεδρίας με την οποία συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά αλλά η κυρία Παλιαδέλη θα ολοκληρώσει αυτήν την έκθεση έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ένα πρώτο επιτυχημένο σχέδιο. Επίσης, επιθυμώ να σας υπενθυμίσω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ε, στείλουμε μία αντιπροσωπεία μας ε, στην Βασλάβ. Ε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πω Μπρέσλα, αλλά δεν είναι Μπρέσλα, είναι Βασλάβ. Κατόπιν τούτου θέλω απλώ να προσθέσω ότι και η δική μου πολιτική ομάδα συμπτωματικά θα βρίσκεται εκεί με το Προεδρείο. θα υπάρχουν και άλλες συνεδριάσεις, All for Europe και πολλές άλλες εκδηλώσεις και ο Μπόρις βεβαίως χαίρεται πάρα πολύ γιατί αυτή είναι η γενέτειρά του. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας ε, θα έχουμε ενδεχομένω να κάνουμε και με το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Με μεγάλη αγωνία περιμένουμε τις ε, νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νέα προγράμματα, εκπαίδευση, αθλητισμός νεολαία. Θα υπάρξουν πολλές και ζωντανές συζητήσεις γιατί όλες οι απόψεις που ακούσαμε είναι αντίθετες με αυτό ε, το οποίο είχαμε διακηρύξει πριν από δύο χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε αυτή τη σύγκρουση και ελπίζω να μας υποστηρίξετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω ε, τι ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Θα δώσω τη δυνατότητα στους υπουργούς ε, να μιλήσουν για όχι περισσότερο από 15 λεπτά. Θα μας πούν τι ελπίζουν να δρομολογήσουν τους επόμενους 6 μήνες γιατί απλά για δρομολόγηση θα πρόκειται. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει ούτε τον κόσμο ούτε το Συμβούλιο. Απλά μπορεί κανείς να συνεχίσει αυτά τα οποία έχουν ήδη αρχίσει άλλοι και να παραδώσει τη σκητάλη στην επόμενη Προεδρία. Και από ό,τι είδα κάνετε κι εσείς ε, ό,τι κάνουν και οι ε, προηγούμενες ε, κυβερνήσεις, δηλαδή δουλεύετε στο πλαίσιο αυτό της Τρόικας του Προκατόχου, του Ενεργού, Προέδρου ή οτιδήποτε άλλο και του Διαδόχου. Ξεκινάμε λοιπόν με την Υπουργό ε, παιδείας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Χολ. Ε, παρακαλώ κύριε Χολ, έχετε το λόγο. E, κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτέ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, για πρώτη φορά η Πολωνία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης. Για μας είναι κάτι το τελείως καινούριο και οι συναντήσεις μας μαζί, σου, μαζί σας ε, είναι για μας σαν μάθημα. Αισθανόμαστε σαν μαθητές στα πλαίσια μιας διαβίου μάθησης ή σαν να είμαι μπροστά σε εξεταστική επιτροπή. Η συνεργασία βέβαια είναι κάτι το οποίο μας εξάπτει επίσης και αυτά που μάθαμε από τη δραστηριότητα των δύο προηγουμένων προεδριών είναι κάτι που μας βοήθησε πολύ. Τις ευχαριστώ για τις συμβουλές που μας χορήγησαν. Γιατί είναι κάτι που με βοήθησε πολύ να προετοιμαστώ για τους επόμενους έξι μήνες, για την Προεδρία μας δηλαδή, και θέλουμε να επιδείξουμε την ίδια αλληλεγγύη. Την, αλληλεγγύη που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην Πολωνία το 80 με 89. Αλληλεγγύη που αφορά και τις γειτονικές μας χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική του 2020 δείχνει ότι η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί με βιώσιμο και ευφυή τρόπο με χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό και με περισσότερη απασχόληση και καινούρια είδη θέσεων απασχόλησης. Η Παιδεία και η νεολαία φυσικά είναι πολύ σημαντικές προτεραιότητες. Ειδικά για τη νεολαία η Πολωνική Προεδρία θέλει να διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης γιατί εδώ αρχίζει μια νέα φάση διαλόγου και συνεργασίας 18 μήνυ Η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία μας έδωσαν μαθήματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε, που ήταν πολύτιμα για μας και συμβουλές. Η Πολωνική Προεδρία θα βασιστεί κυρίως στην νεολαία και την παιδεία, όπως λέει και το ψήφισμα ή τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συνεργασία μέχρι το 2018. Ε, άλλο από τα κύρια θέματα της Προεδρίας μας θα είναι η ενδυνάμωση και προώθηση των ευκαιριών και ανταλλαγών που πρέπει να έχουν οι νέοι από ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και από τις ανατολικές χώρες και τον Κάφκασο. Να υπάρξει διάλογος και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ χωρών ως προς την νεολαία. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση και για περαιτέρω συγκλήσεις των χωρών αυτών με την Ένωση. Η ανατολική διάσταση της κινητικότητας είναι αντικείμενο μιας ανακοίνωσής μας που λέει ότι με την ενδυνάμωση των προσωπικών επαφών και της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και θεσμών μπορούμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών και σε χώρες γειτονικέ μας ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και να δημιουργηθεί μια ανοιχτή κοινωνία έτοιμη για συνεργασία. Σχεδιάζουμε το Συμβούλιο για την Νεολαία και τον Αθλητισμό να καταλήξει στα συμπαράσματά του για την ανατολική αυτή διάσταση των προβλημάτων κινητικότητας και νεολαίας και θα θέλαμε όλες οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα συνεργασίας μεταξύ νέων. Το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Για μας είναι μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες των πολιτών στην Ευρώπη είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνία των πολιτών, για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το σημαντικό εδώ είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι νέοι είναι οι πιο ενεργοί για τον εθελοντισμό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι η εφαρμογή της στρατηγικής του 2020 και του στρατηγικού πλαισίου για την παιδεία βασίζεται σε δύο προτεραιότητες. Τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων και σήμερα ο συνάδελφός μου εδώ από την κυβέρνηση, η καθηγήτρια Κουντρίτσκα, που είναι υπουργό Παιδείας, θα σας μιλήσει για το θέμα αυτό και η άλλη προτεραιότητα εκπαίδευση για κινητικότητα. Οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και οι νέοι, πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που διαθέτουν για μεγαλύτερη κινητικότητα και επαγγελματικά και εκπαιδευτικά αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν από από μικρή ηλικία. Έτσι θα αποφευχθούν οι δημιουργίες κοινωνικών ανισοτήτων και τονίζω ιδιαίτερα τη σημασία του προγράμματος Κομίνιους... που αφορά εκπαιδευτικά ιδρύματα α, για παιδιά και μικρής ηλικίας από τον υπηαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο. Το πρόγραμμα αυτό δίνει ευκαιρίες στους μαθητές ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που διαθέτουν για κινητικότητα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά επαναλαμβάνω. Μία άλλη πρωτοβουλία που λέγεται Youth on the Move υποστηρίζει το στόχο κάθε Ευρωπαίος και Ευρωπαία να έχει τη δυνατότητα να μορφωθεί σε χώρα άλλη από τη δική του. Το Συμβούλιο έχει τονίσει πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα ως προς την εκμάθηση γλωσσών, την γλωσσομάθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης στο ψήφισμά του για την πολυγλωσσία παρόμοια θέση πήρε και η Πολωνική Προεδρία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για γλωσσομάθεια που είναι σημαντικές για την κινητικότητα αυτή, την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα. Η γλωσσομάθεια είναι βασικός παράγων για την οικονομική ανάπτυξη πλέον και για τη μελλοντική απασχόληση των νέων. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να, να προωθηθεί η γλωσσομάθεια ιδιαίτερα για γλώσσες λιγότερο χρησιμοποιούμενες. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνει κανείς τη γλώσσα της γειτονικής χώρας. Τα παιδιά να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα όσο το δυνατόν νωρίτερα. Παραδείγματο χάρη τα γλωσσικά μαθήματα να αρχίζουν από το δημοτικό. Ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνεργασία και εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η Προεδρία επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη γλωσσομάθεια για να υποστηριχθεί η κινητικότητα. Το Νοέμβριο σχεδιάζουμε να εκδοθούν αυτά τα συμπεράσματα για την εκπαιδευτική ιδιαίτερα κινητικότητα θα οργανωθούν διασκέψεις στη Βαρσοβία από την Προεδρία και τα γλωσσικά προσόντα θα θεωρούνται σαν μία από τις βάσεις για την επαγγελματική επιτυχία στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο θα οργανωθεί μια τέτοια διάσκεψη και τον Οκτώβριο. Θέμα θα είναι η κινητικότητα από τους νέους μέχρι και τους πιο ηλικιωμένους πολίτες. Επίσης προτείναμε να οργανωθεί διάσκεψη το Οκτώβριο στο Γκτάνσκ για την διαβίου μάθηση για καλύτερη αποσχολησιμότητα. Άλλο θέμα είναι οι διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων και η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόκτησης προσόντων. Κυρίες και κύριοι, η Πολωνική Προεδρία θέλει επίσης να ασχοληθεί με το θέμα της διαβίου μάθησης και της συμμετοχής των ενηλίκων σε μαθήματα στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Είναι ουσιαστικό να μπορούν και αυτοί έτσι να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους και μία ενεργή ζωή στον πολιτικό, στο στίβο της κοινωνίας. Η συμμετοχή λοιπόν και των ενηλίκων στην εκμάθηση για καλύτερη για απόκτηση περισσότερων προσόντων. Ακόμα και άτυπη εκπαίδευση να χρησιμοποιηθούν δηλαδή περισσότερο τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του προγράμματος Grunding. Σκοπεύουμε να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα ή ανακοίνωση του Συμβουλίου τον Νοέμβριο για αυτά. Κυρίες και κύριοι, τον Ιούνιο η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση για το πολιετές ε, δημοσιονομικό της πρόγραμμα το οποίο θα αναλυθεί εις βάθος από την Προεδρία και στα τέλη του έτους θα υποβληθούν συγκεκριμένα προγράμματα μέχρι το 2020 για την παιδεία και την νεολαία. Καλό θα ήταν τα προγράμματα αυτά να αφορούν περισσότερο την στρατηγική του 2020 Πρέπει να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και η προώθηση των ευρωπαϊκών ιδεοδών μεταξύ των Ευρωπαίων μέσω της πολιτισμικότητας και της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη. Πριν να μπει στην Ένωση η Πολωνία ήμουν διευθύντρια ενός σχολείου και συμμετείχα σε προγράμματα νεολαίας όπως το Σόκρατες και θυμάμαι ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον για τους μαθητές αλλά και για τους δασκάλους η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα γιατί μάθαμε πολλά για τα τελωνία ας πούμε, για διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών, για τα ήθη και έθιμα των χωρών και αποκτήσαμε καινούριου φίλους και εμπειρίες έγιναν ανταλλαγές και οι μαθητές που πήγαιναν στις ανταλλαγές αυτές γίνονταν σαν πρεσβευτές της Ένωσης. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι χάρη στη συμμετοχή των μαθητών και φοιτητών σε αυτά τα προγράμματα ανταλλαγής είπε ναι τελικά η Πολωνία σε μεγάλη πλειοψηφία για την ένταξή της στην Ένωση διότι οι νέοι ήξεραν τι είναι ένωση και ήθελαν να, συμμετέχουν αυτήν, να συμμετάσχουν σε αυτήν. Επίσης χάρη στα προγράμματα ανταλλαγών ιδιαίτερα με τους ανατολικούς μας γείτονες θέλουμε και πάλι να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους πρεσβευτές της Ένωσης σε εισαγωγικά. Γιατί και εκείνοι έτσι μπορούν μια μέρα να αποφασίσουν να ενταχθούν, γι' αυτό τέτοιου είδους προγράμματα ανταλλαγής καθηγητών, διδασκάλων, μαθητών και φοιτητών είναι κάτι το πολύ χρήσιμο. Όλα αυτά σας τα λέω με βάση προσωπικές εμπειρίες. Κυρία μου, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας παρουσίασα τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασίας του Συμβουλίου ως προς τα θέματα της παιδείας και της νεολαίας για το επόμενο εξάμεινο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα πετύχουμε αυτούς τους στόχους και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε στενά με όλες τις χώρες της Ένωσης και σας προσκαλώ όλους να συμμετάσχετε και εσείς στις εκδηλώσεις που θα οργανώσουμε ως Προεδρία. Ευχαριστώ δε για την προσοχή σας και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις ή απορίες. Äh, Έχω λοιπόν μια σειρά συναδέλφων που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα όμως ε, να σας επισημάνω το εξής, ότι σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ε, όπου ε, εμφανίζονται αλλαγές στα προγράμματα τα οποία έχει μαγειρέψει η Κομισιόν σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο εσείς αναλαμβάνετε τα ενία. Ε, χτες είχα τη χαρά να συζητήσω με εκπροσώπους της Επιτροπής οι οποίοι μου εξήγησαν ε, ποια ακριβώς μορφή θα λάβουν τα νέα προγράμματα. Και αν κατάλαβα καλά ε, δεν θα υπάρχει πλέον πρόγραμμα Κομένιους, τουλάχιστον με αυτό το όνομα. Δεν θα υπάρχει πρόγραμμα με το όνομα Κομμένους Ρέγγιο, το οποίο σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Χάνεται λοιπόν ε, ένα σήμα, αν θέλετε. Και όταν έχει ε, καταξιωθεί ένα σήμα, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το ακυρώνουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι ιδιαίτερα για τον τομέα ε, της ε, εκπαίδευσης ε, και του πολιτισμού η Κομισιόν ε, σκέπτεται να αυξήσει σημαντικά τα κονδύλια χρηματοδότησης. Όμως όσο δεν γνωρίζω τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτό το μαύρο κουτί, λέει η Πρόεδρος, είναι πολύ δύσκολο να χειροκροτήσουμε. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώς τι, πώς, τι, γιατί, ποιον, σε ποιον θα δοθούν χρήματα ποιο είναι το ποσοστό που θα εκταμιευτεί για το Κομένιους, ε, για το Εράσμους, για το Λεωνάρντο, για την νεολαία, για τον αθλητισμό. Όσο δεν γνωρίζω αυτά τα ποσοστά δεν μπορώ να χειροκροτήσω με την καρδιά μου. Φοβάμαι λοιπόν και γι' αυτό το λέω ευθύ εξ αρχή ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο πριν από δύο χρόνια απορρίψαμε κατηγορηματικά, δηλαδή να έχουμε το ίδιο πρόγραμμα με νέο όνομα Use on the Move, αυτό ε, αποσύρθηκε και τώρα επανέρχονται και λένε θα υπάρχει εράσμους για όλους ή κάτι παρεμφερές. Διερωτώ λοιπόν και παρακαλώ να γίνετε κι εσείς δικηγόρος της Επιτροπής δικηγόρος λοιπόν της Επιτροπής, με γιατί το πρόγραμμα δεν μπορεί να ε, εξακολουθεί να ονομάζεται διαβίου μάθηση και στο πρόγραμμα αυτό να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν επάνω, να υπάρχουν οι οριζόντιες παρεμβάσεις και μέσα στο πρόγραμμα να υπάρχει το Εράσμους, το Κομένιους, ε, ένας άλλος ε, πυλώνας που θα αφορά τη νεολαία. Γιατί λοιπόν να πρέπει να ανακαλύψουμε ένα νέο όνομα και παρακαλώ εκ βάθους καρδίας την Προεδρία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Ε, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι αυτό το επιθυμεί το Συμβούλιο και έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Ε, κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά την Πολωνική Προεδρία να κάνει λογικά πράγματα. Όταν λέτε ότι εγκρίθηκε ε, το πρόγραμμα Κομένιους ότι εντωμεταξύ είναι ένα γνωστό πρόγραμμα, είναι σήμα όπως το χαρακτήρισα, όχι τόσο όσο το Εράσμους, γιατί το Εράσμους δρομολογήθηκε το 87. Έχει όμως και αυτό το Κομένιους ένα όνομα γνωστό. Γιατί να, το, να εξαφανιστεί και οι άνθρωποι να λένε «Α, χάθηκε πια αυτό το πρόγραμμα». Αυτή λοιπόν είναι η έκκληση ε, που απευθύνω στην Πολωνική Προεδρία να μην μας εγκαταλείψει στον αγώνα μας ε, και η Κομισιόν πριν καταθέσει ένα νέο πρόγραμμα, να δει ε, και να διαμορφώσει το νέο πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να το δεχτούμε. Ε, καλωσορίζω τη συνάδελφο από τους ε, σοσιαλδημοκράτες Κάμα Εβέρτ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό για αυτά που μας είπε. Πάρα πολλά από αυτά μπορούμε να τα δεχθούμε στην Επιτροπή μας με κλειστά τα μάτια <clears throat> και σας ευχόμαστε καλή τύχη στο ιδιαίτερο φιλόδοξο πρόγραμμα ε, το οποίο ε, σκοπεύετε να ε, εφαρμόσετε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Πακ. Κοιτάξτε, όλα αυτά μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Νομίζω ότι βεβαίως και χαιρόμαστε όλοι για το ότι η Κομισιόν μας ανακοίνησε ότι προτίθεται να αυξήσει σημαντικά ε, τα κονδύλια ε, στον προπλογισμό για τον πολιτισμό. Όμως οι ανησυχίες της κυρίας Πακ ότι πράγματι ως Επιτροπή ε, έχουμε ανησυχίες ότι σε τελική ανάλυση αυτά τα ιδιαίτερα προγράμματα που είχαμε κάπως θα ε, χατούν, ε, δεν θα είναι εμφανή ε, και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορούμε να δώσουμε κατευθύνσεις. Θα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλος τομέας πολιτισμού που χρηματοδοτείται αφιδός, αλλά δεν θα ξέρουμε πού ακριβώς διοχετεύονται τα κονδύλια και δεν θα ξέρουμε και το ακριβές περιεχόμενο των προγραμμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και <clears throat> θέλω να σας πω δεν καταλαβαίνω γιατί επιτυχημένα σήματα όπως τα χαρακτηρίσαμε στον τομέα του πολιτισμού γιατί να πρέπει αυτά να εγκαταλειφθούν προς όφελος άλλων όπου οι άνθρωποι πρέπει καταρχήν να συνηθίσουν ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό ε, που παλαιότερα ήταν το Erasmus, το Comenius, το Youth in Action. Όλα αυτά πραγματικά είναι ανησυχία, είναι, είναι ανοησία. Είναι ανοησία τα επιτυχημένα προγράμματα να τα εγκαταλείψουμε και να εφεύρουμε νέα ονόματα ή όλα να μπουν στην ίδια δεξαμενή. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω και εγώ να προσπαθήσετε και εσείς ε, στο Συμβούλιο τα προγράμματα τα οποία κατά το παρελθόν αποδείχτηκαν επιτυχημένα να επανέλθουν, να μπορεί κανείς να τα αναγνωρίσει και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι έχουμε αυτό ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα Youth in Action ε, που αφορά κυρίως την άτυπη εκπαίδευση. Νομίζω λοιπόν ότι πέρα από το ότι βεβαίως ε, και επιθυμούμε να εκπαιδεύουμε σωστά τους ε, νέους και τα παιδιά να τους προετοιμάζουμε για, το, για την επαγγελματική τους ανασχόληση άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει κινητικότητα όμως αυτά όλα σωστά όμως τον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης όπου το θέμα δεν είναι τόσο να έχουμε κάτι άμεσο και απτό για το αποτέλεσμα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι απλά η διαπολιτισμική μάθηση, να γνωριστούν οι, νέες, οι νέοι μεταξύ τους, να αποκομίσουν εμπειρία στο εξωτερικό, να βρεθούν με νέους από άλλες, ε, από άλλα κράτη να περάσουν ένα χρονικό διάστημα μαζί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει τόσο υψηλή αξία που δεν μπορεί κανείς ε, να την εκφράσει με σχολικούς βαθμούς και νομίζω ότι αυτό είναι εξίσου σημαντικό όσο και η καθιερωμένη, η τυπική εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πολύ αυτόν τον τομέα της ε, άτυπης εκπαίδευσης ε, να μην τον εντάξετε στους καλούς στόχους του 2020 αλλά να ε, τον αφήσετε να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια παράκληση που πρέπει να τη μεταφέρετε στο Συμβούλιο Υπουργών. Βεβαίω και είναι πολύ ωραίο να έχουμε περισσότερα κονδύλια για την παιδεία και τον πολιτισμό. Ξέρουμε όμως από την εμπειρία μας ότι ιδιαίτερα το Συμβούλιο Υπουργών είναι εκείνο που πολύ χαρά βαίνει σε περικοπές. Ε, θερμότατη λοιπόν παράκληση προς εσάς ε, που θα είστε προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας να μεριμνήσετε κι εσείς έτσι ώστε αυτά τα οποία πρότεινε η Κομισιόν την αύξηση κοντιλίων να μην το ακυρώσει το Συμβούλιο Υπουργών. Και σας παρακαλώ επίσης ε, τα καλά σήματα, τα επιτυχημένα προγράμματα να τα διατηρήσετε για να μπορούμε με αυτά να προβάλλουμε και στο μέλλον την Ευρώπη. ο κ. Φίσας η ε, Αεξέλα. Με ανησύχησε λίγο αυτό που είπε η κυρία Πακ για την αλλαγή των ονομάτων Κομένιους, Εράσμους κλπ. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Εράσμους έχει κάνει για την Ευρώπη πολύ περισσότερα από ότι πολλές συνθήκες. Είναι πολύ δημοφιλές Οπότε είναι κρίμα να χαθεί αυτό το σύμβολο με αλλαγή ονόματος. Συνεπώ θα ζητούσα από την Υπουργό να επιμείνει να διατηρηθούν τα πράγματα που έχουν γίνει καλά, που έχουν γίνει σωστά. Ε, γιατί στην πολιτική πολύ συχνά ο καινούριο θέλει να τα αλλάξει όλα, όλα τα προηγούμενα, είτε είναι καλά είτε κακά. Μαζί με τα, χλωρά, με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Ε, Εγώ ε, για το θέμα το, του αθλητισμού ε, και γνωρίζω πολύ καλά επίσης πόσο σημαντική, σημαντικός είναι ο εθελοντισμός. Χωρίς τον εθελοντισμό ο αθλητισμός δεν θα υπήρχε. Ε, ο εθελοντισμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικός ε, και θα πρέπει οι εθελοντές να λαμβάνουν κατάρτιση. Επίσης η εκπαίδευση της γλώσσας είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να μαθαίνουμε τις γλώσσες τουλάχιστον των γειτονικών μας χωρών ακριβώς ε, για να αυξήσουμε και την κινητικότητα. Ε, και δεν θα πρέπει να μαθαίνουμε μόνο τα αγγλικά. Ε, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πάμε να δουλέψουμε ή θα πάνε να δουλέψουν οι νέοι. Δυστυχώς δεν άκουσα να μιλάτε καθόλου στην παρουσία σας για την επαγγελματική κατάρτιση. Για μένα η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική σήμερα. Έχουμε ίσως πολλούς πτυχιούχους πανεπιστημίου, δεν έχουμε όμως αρκετούς επαγγελματίες σωστά καταρτισμένους ε, και θέλουμε το στάτους της επαγγελματικής κατάρτισης ε, να ε, αυξηθεί, να βελτιωθεί. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφος Μπόρις έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που παρουσιάσατε τις πολωνικές ε, προτεραιότητες. Η ερώτησή μου αφορά την οριζόντια προσέγγιση. Έχουμε υιοθετήσει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 που αποτελεί την πολιτική μας ατζέντα για τις αλλαγές τα επόμενα χρόνια και είναι και μια απάντηση στην κρίση μέσω της εφιούς ανάπτυξης ε, ε, ε, και ε, υποστηρίζεται πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν. Με, στις συναντήσεις σας με τους υπουργούς στο Σύμβουλο Υπουργών θα ε, προωθήσετε τους στόχους της ε, ατζέντα αυτής της Ευρώπης 2020 έτσι ώστε ε, να υλοποιήσουμε πραγματικά ε, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ε, εφαρμογή της στατικής Λισαβόνας. Δηλαδή θα προσπαθήσετε να πείσετε τους υπουργούς ότι είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες. Χωρίς την συμμετοχή των κρατών μελών κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Δεύτερον, συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι σε όλα τα κοινοτικά προγράμματα χρειαζόμαστε ε, μια σοφή εξέλιξη, όχι μια επανάσταση. Συνεπώς, ε, όταν ε, εργαστείτε στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, θα πρέπει να δώσετε σημασία και στα προγράμματα συνοχής έτσι ώστε από τα 370 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για τις πιο αδύναμες περιοχές ε, να δοθεί ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό στην εκπαίδευση μέσα στην στρατηγική ατζέντα Ευρώπη 2020. Ähm, Κύριε Μακλάρκεν, Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας του προγράμματος της Προεδρίας με, βάση, με ιδιαίτερη έμφαση στην νεολαία και την παιδεία. Και, μας, και εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορούμε να ακούσουμε τους νέους και μας ενδιέφερε ιδιαίτερα η ιδέα σας για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και μάλιστα είμαι εισηγήτρια για το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων και για, και για μας σημαντικό να μπορέσουν οι νέοι να εκμεταλλευτούν το δικαίωμα της κινητικότητας που έχουν. Θα παρακολουθήσω λοιπόν κατά πόσον η Προεδρία σας θα εφαρμόσει τους στόχους αυτούς ώστε να μπορεί κανείς να ασκήσει το επάγγελμά του σε πολλές χώρες και όχι μόνο στη δική του το Δεκέμβριο και εμείς θα εγκρίνουμε μια σχετική έκθεση και θα εκμεταλλευτούμε και τις δικές σας προτάσεις. Έχουμε κι άλλο έναν υπουργό, ε, η επόμενη κυρία, ε, που θα μιλήσει για την ανώτατη εκπαίδευση. Καλύτερα να περιοριστούμε ε, στα θέματα που αφορούν την υπουργό που μας έχει ήδη μιλήσει. Επόμενος ομιλητής, Τάκουλα. Κυρία... Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό που μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Και από ό,τι φαίνεται η Πολωνική Προεδρία μας υπόσχεται περισσότερα κονδύλια στα θέματα εκπαίδευσης, ε, παιδείας και πολιτισμού. Τα προγράμματα για την ε, παιδεία έχουν στεφθεί από επιτυχία και πρέπει να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά. Και η Πολωνική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την εξέλιξη των προγραμμάτων έτσι ώστε να γίνουν ακόμα πιο πετυχημένα. Γιατί είναι αλήθεια πως εξετάζοντας τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης βλέπουμε πως μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Άκουσα τι είπαν και οι συνάδελφοι για το θέμα της μάρκας. Ε, η, στη Φιλανδία λέμε μερικές ε, φορές ε, δεν πρέπει ποτέ να αλλάζουμε κάτι το οποίο δουλεύει. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε. Εγώ θα προτιμούσα να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα προγράμματα. Το Εράσμους ήταν μεγάλη επιτυχία, όπως και να το κρίνουμε. Πιο σημαντικό βέβαια από το όνομα είναι το περιεχόμενο. Πώς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια ευρωπαϊκή αξία σε αυτά τα προγράμματα και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα Εράσμους για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ε, για παράδειγμα, ε, δεν πρέπει να ανατρέφουμε τα παιδιά μας με στόχο απλώς να αυξήσουμε το ΑΕΠ της χώρας μας. Η παιδεία έτσι κι αλλιώς είναι εθνική ε, υποχρέωση και εθνική αρμοδιότητα, αλλά ας δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την κατάρτιση με τις ε, ανάγκες αγοράς έτσι ώστε να ε, έχουμε εργατικό δυναμικό ποιοτικό καταρτισμένο και όχι μόνο εργατικό δυναμικό και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι επαρκώς καταρτισμένοι. Η Πολωνία κατά διάρκεια της Προεδρίας της ε, ελπίζω ότι θα προωθήσει και την ποιότητα της κατάρτισης των εκπαιδευτών. Η ε, μελέτη PISA μας δείχνει ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Αν θέλουμε να βελτιωθεί η παιδεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξ ονόματος των ε, φιλελευθέρων, ε, εύχομαι καλή πτυχία στην Πολωνική Προεδρία και παραλαμβάνω ότι το σημαντικό είναι το περιεχόμενο. Ας ε, αφιερώσουμε τις προσπάθειές μας στο περιεχόμενο. Ανεξάρτητα από το φιαλίδιο στο οποίο κλείνουμε το περιεχόμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κουρία. Ε, κύριε Υπουργέ, θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει από όλους τους ε, συναντέλφους, ε, ξεκινώντας από την Πρόεδρο, το είπε και αυτή. Το επαναλαμβάνω όμως και εγώ για να καταλάβετε ότι αυτή η διάθεση που υπάρχει να προστατευτούν τα πολιτικά προγράμματα για τους νέους, για την εκπαίδευση, αυτό είναι κάτι που ε, μας απασχολεί όλους, ε, βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας, ε, διαπολιτικά, διατομεακά. Εγώ μιλώ εξ ονόματος του ΕΛ, αλλά και οι σοσιαλιστές και όλοι οι άλλοι, όχι έτσι γενικά και ορίστα, όλοι μας λοιπόν επιθυμούμε αυτά που προτείνει η Κομισιόν να αναθεωρηθούν. Γιατί μέσα από αυτά τα προγράμματα μας δόθηκε ευκαιρία η Ευρώπη να αντιμετωπίζεται ως ένας σοβαρός συνομιλητής, να αποκτήσει σοβαρότητα μέσα από τη διάρκεια των ετών. Εμείς ε, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρώπη όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα προγράμματα βοήθησαν στο να υπάρχει μια πραγματική ευαισθησία στα κράτη-μέλη και γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρούμε ότι ε, τουλάχιστον ε, αυτά τα προγράμματα να αποτελέσουν ε, ε, βάση συνεργασίας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα οποία είπατε για τους νέους, διότι πράγματι οι νέοι αποτελούν μια κατηγορία στην οποία πρέπει να παρέμβουμε για το μέλλον της Ευρώπης εσείς ε, θα ολοκληρώσετε ε, την πρωτεύουσα του 2011 που είναι το έτος ε, της εθελοντικής εργασίας. Αυτό το θέμα είναι βέβαια εθνικής αρμοδιότητας. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει ένα βήμα περαιτέρω για να δείξει ότι πράγματι ενδιαφέρεται και αυτό το θέμα και μπορεί να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σε ευχαριστώ καταρχήν γιατί παρουσιάσατε ιδιαίτερα εύγλωτα τις προτεραιότητές σας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ε, πρόσφατα υπήρξε ένα συνέδριο με θέμα ε, κατά πόσον ε, μπορεί να υπάρχει κινητικότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς έχετε διερωτηθεί με το πώς ε, μπορούν οι νέοι στην Ανατολική Ευρώπη να είναι περισσότερο κινητικοί. Αναφέρομαι, όπως σας είπα, στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Ε, πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Ε, κατόπιν τούτου τέτησαν όλες οι ερωτήσεις. Πλάστα σε αυτό το γύρο. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις που κάνατε, οι οποίες παρατηρήσεις σίγουρα θα με βοηθήσουν στη δουλειά μου. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στη συζήτηση ε, που διεξάγεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σχετικά με τα προγράμματα. Γνωρίζουμε ότι τα προγράμματα αυτά θα συνεχιστούν, ε, επίσης θα συνεχίσουν ε, να χρηματοδοτούνται. Το θέμα βέβαια είναι πώς, με ποιο τρόπο. Αναμφίβολα αυτό θα είναι το θέμα πολλών ε, συζητήσεων και αναλύσεων που θα ακολουθήσουν. Αυτό μπορώ να το πω ήδη σήμερα. Εγώ προσωπικά ε, θυμάμαι και άλλα ε, προγράμματα κατά παρελθόν που σήμερα δεν υπάρχουν. Σήμερα υπάρχει το Σοκράτης, Σοκράτης το Κομένιους, αλλά παλαιότερα υπήρχαν και άλλα. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να διατηρηθούν αυτά τα προγράμματα ακόμα και εκείνα που αφορούν ε, τα μικρά παιδιά, ε, την προσχολική ε, ηλικία, η εκμάθηση ξένας γλώσσας. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση της κινητικότητας. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδου ε, προγράμματα που όπως σας είπα αφορούν τα πολύ μικρά παιδιά, τους νέους προσχολικής ε, ηλικίας γιατί μέσα από αυτά τα προγράμματα συμβάλλουμε και στην ιδέα της ε, συνοχής. Η κυρία Πάκα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, έχοντας βέβαια κατά νου το πρόγραμμα Comenius και κάποια άλλη κυρία προλαλήσασα που δεν συγκράτησα το όνομά της αλλά και εκείνη ε, αναφέρθηκε ε, σε αυτά τα προγράμματα. Ελπίζω μέχρι το τέλος της ε, Προεδρίας να μπορώ να συγκρατήσω το όνομά σας. Πάντως θέλω να σας πω ότι κάνετε θαυμάσιες παρατηρήσεις για τα προγράμματα αυτά. Και ο κύριος Τάκουλα και εκείνος είπε πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα αυτά, την αξία που προσφέρουν. Ίσως ε, το θέμα να μην είναι τόσο σημαντικό το θέμα του ονόματος, αλλά το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ίσως αυτό να είναι σημαντικότερο. Είναι λοιπόν ε, ουσιώδες το ε, να προσφέρουμε στους φοιτητές, στους νέους, στις οργανώσεις νέων τη δυνατότητα να εργαστούν, να συνεργαστούν με γειτονικέ χώρες της Ευρώπης, κυρίως ε, με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η κυρία Μακλάκεν μίλησε για την κινητικότητα των νέων. Το πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την κινητικότητα των νέων. Επίσης αναφέρθηκε από τον τελευταίο μιλητή ότι η ανατολική διάσταση της κινητικότητας, δηλαδή το να υπάρχει κινητικότητα στην Ανατολική Ευρώπη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι οι νέοι θα είναι περισσότερο κινητικοί ε, εάν ε, ενισχύσουμε οικονομικά τις οργανώσεις τους. Και αυτό ελέγχθη και κατά τη διάρκεια ε, του συνεδρίου που χώρα με θέμα την ε, κινητικότητα των νέων στην Ανατολική Ευρώπη. Κατόπιν το θέμα σχετικά με την ε, διαδικασία της Μπολόνια. Εκεί νομίζω μπορούμε να μην βαθύνουμε περαιτέρω. Εσείς αναφερθήκατε στο ότι η διαβίου μάθηση είναι σημαντική και το ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ε, εκπαίδευση, την περαιτέρω κατάρτιση των ενηλίκων. Έγινε λόγος για την επαγγελματική κατάρτιση. Είπατε ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα σημαντικό θέμα. Ε, και έχετε δίκιο. Εμείς επιθυμούμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η επαγγελματική κατάρτιση να αντιμετωπιστεί θετικά, να ενισχύεται, να προωθείται στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποκτούν περισσότερα επαγγελματικά προσόντα να συνεχίζεται διαβίου η επαγγελματική κατάρτιση. Θεωρώ ότι έχει σημασία το να μπορεί κανείς ε, να αποκτά ε, προσόντα, ε, μάλιστα όχι με καθαρά τυπικό τρόπο. Και επ' αυτού θα κάνουμε συζητήσεις και θα ανταλλάξουμε εμπειρίες. υπόθηκε το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προσόντα ε, και πώς μπορούμε να ε, έχουμε καλύτερη εμπειρία. Ο κύριος Μπόρις ε, έθεσε ένα ερώτημα που αφορά στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Ετέθη επιτάπητο στο θέμα της συνοχής. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη, η στρατηγική Ευρώπη 2020, η στρατηγική αυτή μας προσφέρει συγκεκριμένους δείκτες Αυτούς τους δείκτες προσπαθούν να τους λάβουν υπόψη τους τα κράτη-μέλη και να τους εντάξουν στην εφαρμογή της πολιτικής τους. Με αυτά λοιπόν τα προγράμματα συνεχής και με τα διαθέσιμα κονδύλια οφείλουμε να επιδιώξουμε τη βελτίωση των δικτών. Χάρη λοιπόν της στρατηγικής, με τη βοήθεια της στρατηγικής 2020 έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη λειτουργία και τα αποτελέσματα που ε, απορρέουν από τη χρήση κοντιλίων. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθοριστική σημασία να προγραμματίσουμε σωστά τη χρήση αυτών των κοντιλίων και μάλιστα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιδιώξουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στο τομέα, στο θέμα της ε, κοινωνικής συνοχής. Και εδώ μπορούν να συμβάλλουν και συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν ε, στους ε, καθηγητές, στα σχολεία, ε, προγράμματα τα οποία προβάλλουν συγκεκριμένα προσόντα, τα οποία μπορούν να αποβούν χρήσιμα για να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Όπως είπα και προηγουμένως, επιθυμούμε να προβάλλουμε περισσότερο αυτά τα προσόντα και δεν αναφέρομαι μόνο στις ξένες γλώσσες αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας, την ε, ικανότητα συνεργασίας με άλλους ε, στο πλαίσιο των ε, κοινών προγραμμάτων. Αναφέρομαι επίσης σε ανταλλαγές με άλλες χώρες και νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε νέους που θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι και θα είναι περισσότερο ε, πρόθυμοι να διεκδικήσουν, να αποκτήσουν αυτά τα επαγγελματικά προσόντα. Κοιτάω λιγάκι τις σημειώσεις μου για τις ερωτήσεις που ετέθησαν για να είμαι σίγουρη ότι δεν ξέχασα τίποτα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρξουν και άλλε ευκαιρίε να συναντηθούμε και να συνεργαστούμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι σίγουρη ότι μπορώ να βασίζομαι στην εμπειρία σας ε, για όλα αυτά τα οποία ανέφερα σχετικά με τα προγράμματά μας. Είμαι στη διάθεσή σας και ελπίζω να μπορέσουμε να ε, συνεργαστούμε στο μέλλον με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Υπουργέ. Από την απάντησή σας ε, συνεπέρανα ότι δεν συμφωνείτε απόλυτα μαζί μας ε, τουλάχιστον όσον αφορά τα νέα προγράμματα. Άρα δηλαδή φοβάμαι ότι ε, στο Συμβούλιο δεν θα έχουμε στεναρή παρουσία και εκπροσώπηση για αυτά που είπαμε. Στάνομαι έτσι λοιπόν λιγάκι μόνη και εγκαταλειμμένη και γι' αυτό σας κάνω έκκληση μην ξεχνάτε ότι εμείς το είχαμε αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα διαβίου μάθηση που καλύπτει τα πάντα. Και αν τώρα ε, σε αυτό το πρόγραμμα μπρέλα μπει και ο αθλητισμός ε, και η νεολαία, πάρα πολύ ωραία, δεν διαφωνώ. Όμως τα σήματα αυτά τα οποία δημιουργούν συνειρμούς, τα είπατε και μόνοι σας, κομμένιους, εράσμους, αυτομάτως προκύπτουν συνειρμοί. Όλοι γνωρίζουν το πρόγραμμα εράσμους και το πρόγραμμα κομμένιους, αν δεν το δολοφονήσουμε, σύντομα θα το γνωρίζουν επίσης όλοι οι πολίτες. Παρακαλώ λοιπόν θερμά να τίνετε ευήκον ους ε, στο Κοινοβούλιο, γιατί εμείς επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτά τα σημαντικά σήματα. Είναι σήματα ταύτισης, ε, και τώρα η Προεδρία λέει μα δεν παίζουν ρόλο τα ονόματα. Μα αγαπητή κυρία Υπουργέ, για μα παίζουν ρόλο τα ονόματα και τα σήματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά να αναθεωρήσετε λιγάκι, να αναθεωρήσετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε το θέμα. Δηλαδή μην πάτε στο Συμβούλιο και πείτε δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματα. Εγώ σας λέω, εμάς μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν και πολύ μάλιστα. Παρακαλώ λοιπόν να το λάβετε υπόψη σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το θέμα της ε, συνεργασίας ε, με τα κράτη-μέλη, ε, το θέμα αυτό το εντάσσεται ε, και στο πλαίσιο της ε, πολιτικής γειτονίας δεν έχει σημασία ε, κατά πόσον τα γειτονικά κράτη θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνεργασία μαζί τους. Αυτό έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που ένα από τα βασικά σας θέματα είναι ακριβώς αυτό που σας ανέφερα. και θεωρώ ότι στο πρόσωπό σας έχουμε έναν ε, αμύντορα όλων αυτών των προγραμμάτων αλλά φαντάζομαι καταλάβατε ε, τι ε, θέλουμε να πούμε. Είδα και κάποιους συνεργάτες σας και από το πρόσωπό τους συμπεραίνω ότι πράγματι έπιασαν το νόημα και θα προσπαθήσουν να πείσουν την Κομισιόν ότι ακολουθεί λάθος δρόμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Και θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την επόμενη συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω ε, μια κουβέντα στα όσα είπα προηγουμένως. Προσωπικά ε, ε αξιολογώ ιδιαίτερα το πρόγραμμα Κομένιους και θα ήθελα να συνεχιστούν οι δράσεις του. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω και βασίζομαι στην συνεργασία σας έτσι ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα Κομμένιους. Ελπίζω να με παρεξηγήσατε. Πολύ ωραία, αλλά... Πολύ ωραία, αλλά εμείς δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε αυτά που λέμε και αυτά που επιδιώκουμε μέχρι να τα πετύχουμε. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Κουντρίτσκα, Υπουργός Επιστημών και Ανώτερης Εκπαίδευσης. Έχετε παρακαλώ το λόγο.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 πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει το πρώτο προσχέδιο της νομοθετικής πράξης για την κινητικότητα. Επίσης αναμένουμε μια ανακοίνωση για τον εξυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης. Η, η περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερη διότι ζούμε μια οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση, ενώ ταυτόχρονα οι νέοι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν εμπιστεύονται πολύ τις κυβερνήσεις των χωρών τους και τα όργανα των χωρών τους. Και εξαιτία των διαφορετικών αλλαγών που γίνονται, ε, ιδιαίτερα στην ανώτερη εκπαίδευση των πολλών κρατών μελών, ε, πολλοί νέοι έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Οι προκλήση για το μέλλον είναι λοιπόν πολλές και σημαντικές. Η Πολωνική Προεδρία τις γνωρίζει πολύ καλά. Σας διαβεβαιώ. Άλλα και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις. Δεν είναι μόνο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης. Οπότε ευχαριστώ πολύ για το ψήφισμα το οποίο υιοθετήσατε στις 12 Μαΐου του τρέχοντος έτους για το πρόγραμμα ε, κινητικότητας για τους νέους. Και το ψήφισμα το σχετικό με τις ε, σχέσεις πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο. Νομίζω ότι αυτά τα ψηφίσματα δείχνουν το σωστό δρόμο και εμπνέουν όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο. προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο μέλλον. Η κινητικότητα αναφέρθηκε και από την Πρόεδρο ως ένα από τα πιο βασικά προβλήματα της Προεδρίας. Ας το σχολιάσω λοιπόν και εγώ πρώτο πρώτο, διότι αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Και στο Συμβουλίο Εκπαιδείας και στο Συμβουλίο Ανταγωνιστικότητας η θα συζητηθεί το θέμα της κινητικότητας, γιατί η κινητικότητα ε, βοηθάει και στην εφαρμογή της Στατικής Ευρώπη 2020 και στην ε, ανάπτυξη της ε, καινοτομίας, στη βελτίωση της παιδείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ μαζί σας, Πρόεδρε, ότι ότι είναι καλό να διατηρούμε κάποια σήματα, κάποια σύμβολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύμβολα έχουν προσθέμενη αξία. Και αυτό ισχύει και για τα προγράμματα κινητικότητας όπως το Εράσμους και το Κορνέλιους. Κομένιους, συγγνώμη. Ε, η, η Επιτροπή προετοιμάζει προσχέδια αποφάσεων για την κινητικότητα με πρόθεση να ε, εντάξει σε, ένα, ε, σε μια κοινή βάση πολλά προγράμματα κινητικότητας και να προτείνει μια νέα λύση. Εγώ ως τώρα δεν ξέρω ποια είναι αυτή η καινούρια λύση, αυτή η καινούρια βάση. Δεν έχουμε ακόμα γνώση των τελικών προτάσεων της Κομισιόν, αλλά για τα προγράμματα κινητικότητας σαφέστατα το πεδίο εφαρμογή θα διευρυνθεί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε την προσθέμενη αξία τους. Ε, τα προγράμματα κινητικότητα, ιδιαίτερα τώρα που θα διευρυνθούν, θα συνεισφέρουν ώστε να αυξηθεί η, αλληλο, ε, η εμπιστοσύνη. Θέλουμε λοιπόν να ε, αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του Εράσμους και ταυτόχρονα να συμπεριλάβουμε και τους φοιτητές επί Ξέρω ότι τα συστήματα, τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι οργανωμένα με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη και είναι δύσκολο να τους συμπεριλάβουμε, αλλά είναι στόχος μας να συμπεριληφθούν και οι ε, φοιτητές επιδιδακτορικό. Ε, επίσης, ε, άλλος στόχος είναι να διαβρύνουμε το πρόγραμμα Εράσμους και στις γειτονικές χώρες. Ε, έγινε μια ερώτηση για την ε, πολιτική γειτονία με τις ανατολικές χώρες. Ε, εμείς θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στο ε, βασικό εράσμος, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, Εμείς θέλουμε όμως και οι χώρες της Ανατολικής ε, ε, οι ανατολικές γειτονικές ε, χώρες να συμμετάσχουν στο Εράσμους, όχι στο Εράσμους μόντους, στο Εράσμους. Με καταλαβαίνετε έτσι. Έτσι να έχουν με τη δυνατότητα περισσότεροι φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να έχει την πρόθεση να αυξήσει τον προπολογισμό για να επιτύχει σε αυτούς τους στόχους. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ε, η νέα λύση που θα προτείνει η Κομισιόν θα υιοθετηθεί όπως θα προταθεί από το Συμβούλιο. Στις 20 Ιουλίου θα συζητηθεί το θέμα της κινητικότητας. Ε, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα ε, συνέλθει στην Πολωνία με παρουσία των Υπουργών Παιδείας και θα συζητηθούν αυτές οι προτάσεις. Αν το ζήτημα του ονόματος είναι τόσο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το Συμβούλιο και, το, και την Κομισιόν για να δούμε αν οι προτάσεις ε, θα οδηγήσουν σε μια ε, ριζική αναδόμηση του συστήματος ή αν θα οδηγήσουν σε μια εξέλιξη. Γνωρίζω ότι ε, τα σύμβολα έχουν κερδίσει μια θέση στην καρδιά και στο μυαλό των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω το εξής. Κατά τη διάρκεια της ε, διάσκεψης για την κινητικότητα με τους ανατολικούς γειτονές μας αντιληφθήκαμε πόσο μικρή είναι η εμπλοκή αυτών των χωρών στη βασική δραστηριότητα του Εράσμους μόνο 2 3% των φοιτητών από τις χώρες που εμπίπτουν στην ε, σχέση ανατολικής γειτονίας ε, συμμετείχαν σε προγράμματα Εράσμους από το 2006 και μετά. Πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Θέλουμε να διευρύνουμε την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα και να συμπεριλάβουμε όπως σας είπα, σε μεγαλύτερο βαθμό τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Ε, άλλος μας στόχος είναι ο εξυγχρονισμός του Πανεπιστημίου. Το Σεπτέμβριο θα η Κομισιόν θα δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Τον Οκτώβριο θα διοργανωθεί για το ίδιο θέμα στο Σόποτ στην Πολωνία μια διάσκεψη και το Συμβούλιο θα υιοθετήσει συμπεράσματα για το ζήτημα αυτό και πάλι το Νοέμβριο. Όλες οι δράσεις τις οποίες, αναφέρατε για τον ξεχωρισμό του Πανεπιστημίου είναι σημαντικές. Ήδη τις έχετε συμπεριλάβει σε παλιότερο ψηφισμά σας. Αυτό που χρειάζεται λίγο περισσότερο δούλεμα, λίγο περισσότερη επεξεργασία, είναι να μην ερωτούμε μόνο για τις υποδομές και την ποιότητα στα κράτη-μέλη. Να αλλάξουμε δηλαδή τα σχολικά προγράμματα με βάση τη διαδικασία της Μπολόνια για τις ανάγκες αναγνώρισης. Ε, αλλά να δουλέψουμε και στο θέμα της ποιότητας των εκπαιδευτών και των καθηγητών. Εμείς ε, πρόσφατα μεταρρυθμίσαμε την ανώτατη εκπαίδευση στην Πολωνία και κάποιο είπε ότι είναι πιο δύσκολο να μεταρρυθμίσει κανεί την ανώτατη εκπαίδευση παρά τον τομέα τη εξορρυκτική βιομηχανία. Γιατί πολύ γρήγορα όταν κάποιος προσπαθεί να επιφέρει αλλαγές βρίσκει απέναντί του το εκπαιδευτικό προσωπικό Οπότε είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμοστεί μετά σε εθνικό επίπεδο από κάθε χώρα. Η βοήθεια, η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν πολύ χρήσιμη λοιπόν για τα κράτη-μέλη. Συνεπώς πέραν όσων συμπεριλάβατε στο ψήφισμα συνεργασία με τις επιχειρήσεις, ε, ε, γνωριμία με τους επιχειρηματίες, συνεργασία σε εφαρμοσμένες ε, επιστήμες, χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την δημιουργία καινούριων υπηρεσιών, τεχνολογιών και προϊόντων. Πέρα από αυτές τις προτάσεις λοιπόν του ψηφίσματός σας πρέπει να πάρουμε υπόψη και άλλα πράγματα. Ε, έχουμε πρόβλημα για παράδειγμα εξασφάλισης ε, χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της κρίσης. Μετά τα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να ε, δίνουν προσθέμενη αξία μόνο συνεργαζόμενοι με επιχειρήσεις ή πουλώντας τεχνογνωσία τα πανεπιστήμια έχουν και ένα τρίτο ρόλο να παίξουν. Θα πρέπει να μεταμορφωθούν σε καινοτόμα ιδρύματα που θα συνεργάζονται με τις ε, κοντινές επιχειρήσεις και θα είναι δραστήρια σε όλη τους την περιφέρεια. Και όχι μόνο με επιχειρήσεις αλλά και με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάτι τέτοιο είναι μια σημαντική αλλαγή, διότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμόσουν και την ε, διαβίου μάθηση. Ε, είναι ένα τέλειος καινούριο σύστημα για αυτά. Δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα απλώς να πω ότι Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε στο Συμβούλιο χωρίς συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινοβούλιο και Κομισιόν. Και η συνεργασία μας μαζί σας, η χρήση των ψηφισμάτων ε, τα οποία θετείτε, θα είναι ε, προϋπόθεση για μας χρειαζόμαστε εξυγχρονισμό, χρειαζόμαστε εξυγχρονιστικές αλλαγές στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Μόνο έτσι θα πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Ε, είδαμε τις ε, απεργίες στην ε, Ελλάδα, τις διαμαρτυρίες. Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και κατεβαίνουν στους δρόμους, διαμαρτύρονται, διαδηλώνουν. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων τη σημερινή εποχή. Χρειάζεται να συνεργαστούμε και να πιέσουμε και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Όχι τους πολιτικούς, τον ακαδημαϊκό κόσμο. Πρέπει να πιέσουμε μαζί τον ακαδημαϊκό κόσμο για να πετύχουμε το καθήκον μας. Γιατί αλλιώς οι διαφορετικέ αλλαγές, ε, τη χρηματοδότηση, η κρατική χρηματοδότηση, τα προγράμματα ε, συνοχής ε, και σύγκλησης δεν πρόκειται να πετύχουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. σε μερικά θέματα ανταποκριθήκατε όντως αυτά που πιστεύω και εγώ, σε άλλα όχι. Για τη διαδικασία της Μπολόνιας ας πούμε. Εμείς μιλάμε για συμμετοχή, για πλήρη συμμετοχή των κοινοβουλίων, αλλά ο κόσμος που Αυτοί που δεν σκέφτονται καθόλου ότι χρειάζεται αλλαγή είναι ακριβώ οι ίδιοι οι καθηγητές και αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισαν να επιδεικνύουν την ίδια συμπεριφορά με πριν. Όπως με τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό είναι μια δυσκολία στην αλλαγή, για την αλλαγή της νοοτροπίας τους λοιπόν δεν σκέφτονται την απαραίτητη αλλαγή. Μπορεί μάλιστα να πρόκειται και για υπαναχώρηση και κάτι άλλο ακόμα. Όπως είπα προηγουμένως και το συνάδελφό σας, εμείς θέλουμε να σας στηρίξουμε. Θέλουμε να υπάρξει ένα άνοιγμα προς τις γειτονικέ σας χώρες προς την Ανατολή αλλά και προς τον Νότο και προς τον Νότο, προς την Αφρική. Φυσικά χρειαζόμαστε και χρήματα και υποδομές, αλλά τουλάχιστον για τον πολιτισμό και την παιδεία θέλουμε να προσπαθήσουμε να συμμετάσχουν περισσότεροι σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Για μας είναι σημαντικό νομίζω και για σας το ότι δεν μπορεί όλοι όσοι προέρχονται από κάποια ανατολική χώρα και έχουν κάποιο δίπλωμα να αναγκάζονται μετά ως επάγγελμα να γίνουν ταξιτζίδες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τα προσόντα τους και όσοι είναι στην Ένωση και από την Ουκρανία και την Τινησία. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να ασκήσουν τα προσόντα τους. γιατί υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, ε, τεράστια προσόντα και αναγκάζονται να γίνουν ταξιτζίδες. Μα είναι τρομερά πράγματα αυτά. Τέλος πάντων. Συμφωνούμε εδώ απόλυτα. Είπατε ότι πρέπει να βρεθούν πόροι και χρηματοδότηση για την κινητικότητα. Η Επίτροπος Βασιλείου κατά την τελευταία της επίσκεψη εδώ μας είπε ότι ήθελε να επεξεργαστεί αυτό το θέμα της κινητικότητας για να εκμεταλλευτεί τον αερασμό κτλ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την ομιλία σας. Ε, πράγματι είπατε πάρα πολλά από αυτά που θέλαμε να ακούσουμε και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις. Ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ την Υπουργό για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Καταρχήν να υπογραμμίσω αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως. Ε, μας ενδιαφέρουν τέτοια, αυτά, όλα αυτά τα προγράμματα, το Erasmus, το Erasmus Mundus, το Comenius, λειτουργούν σωστά, δεν πρέπει να αλλάξουμε τα ονόματά τους ε, που αποτελούν σήμα κατά τεθέν. Ακριβώς το αντίθετο θα πρέπει να κάνουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις μάρκες, αυτά τα σήματα. Θα ήθελα να ε, σχολιάσω το εξή μετά τα όσα είπε και η κυρία Πακ. Είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε την αότατη εκπαίδευση στις πραγματικές ανάγκες του σημερινού κόσμου. Ο καλύτερος φίλος μου είναι καθηγητής Λατινικών και δεν θέλω είναι να πω ότι θα πρέπει να καταργήσουμε την δασκαλία των Λατινικών ή των, κλασικε τις Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη έτσι ώστε η εκπαίδευση ε, και τα προγράμματα να προσαρμοστούν στις ανάγκες έτσι ώστε να μην έχουμε πτυχιούχους χωρίς ε, θέση εργασίας, χωρίς απασχόληση στο μέλλον. Να υπενθυμίσω επίσης ότι η Επιτροπή μας έχει την, ε, το πρόγραμμα Marie Curie που είναι υποτροφίες, ερευνητικές υποτροφίες, ε, θα ήθελα να το προσέξουμε και να το αναπτύξουμε. Και όσοι εισηγητής για τον αθλητισμό να πω και το εξής. Ε, η, τα διπλά πτυχία πώς θα μπορούσε, μάλλον η διπλή καριέρα, πώς θα μπορούσαμε να επιτρέψουν στους αθλητές μας να συνδυάσουν την αθλητική τους δραστηριότητα με ε, φίτηση στα πανεπιστήμια. Ε, όχι βέβαια να τους ε, δίνουμε καλούς βαθμούς επειδή απλώς είναι αθλητές αλλά να τους βοηθήσουμε, να τους συνδράμουμε ενδεχομένως ε, με κάποια πρόσθετη ε, με κάποια υποστηρικτική ε, διδασκαλία ή με κάποιο άλλο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν και τις δύο τους ε, επαγγελματικές καριέρες. Ευχαριστώ. Yeah, από, από τη Ρουμανία. με την πρόεδρο κυρία Κυρία Χάλ και τους υπόλοιπους εκπροσώπους από την Πολωνία θα ήθελα να σας ε, κολασορίσω θερμά. Για μας ε, είναι μεγάλη χαρά το ότι σας έχουμε ε, σήμερα εδώ. Εχθές στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακούσαμε επίσης τους συναντέλφους και για μένα ως ε, Ούγγρο της ε, Ρουμανίας είναι πολύ σημαντικό το ότι η Πολωνία συνεχίζει το δυναμισμό με τον οποίο το δυναμισμό τον οποίο επέδειξε η Ουγγαρία κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό όπου ο Πολωνός βασιλιάς ίδρυσε ε, το πρώτο Ουγγρικό Πανεπιστήμιο και εκεί ε, έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι Ουγγρικές-Πολωνικές ε, σχέσεις διαμορφώθηκαν ακριβώς γι' αυτό λόγο πολυθετικά. Μιλώ για το πρώην κομμουνιστικό καθεστώς το Νότς Βάρατ Ιδρύθηκε εκεί επίσης ε, ένα πανεπιστήμιο το οποίο όμως το 59 ο Τσαουσέσκου το έκλεισε. Στο Μάρους Βάσαρ και σε άλλες πόλεις ε, ιδρύθηκαν πανεπιστήμια. Τώρα λοιπόν δυστυχώς ε, αντιμετωπίζουμε κρίση στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι αισθητά τα προβλήματα που κληροδότησε ο κομμουνισμός και μετά από 20 χρόνια δεν έχουμε κατορθώσει να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Ε, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ε, θερμός οπαδός ε, της απόλυτης κινητικότητας γιατί όπως είπε και η κυρία Πακ τελικά οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων μας καταλήγουν να γίνονται οδηγοί ταξί ε, σε αυτή λοιπόν την μετακομμουνιστική κρίση έχουμε πλέον μια κοινωνία η οποία καλείται να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ούτε η Ρουμανία αλλά ούτε και η Ουγγαρία εξελίσσονται σωστά. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στην Πολωνία. Στην Ρουμανία έχουμε δύο εκατομμύρια που μετανάστευσαν μόνιμα, είτε αναζητώντας εργασία, είτε για άλλους λόγους, ε, γιατί ήταν φοιτητέ και θέλησαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλα πανεπιστήμια. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα ε, στα συστήματα της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει να επανέλθει η ισορροπία. Οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές και αυτό πρέπει να εξισορροπηθεί ε, προς όφελος των νέων ε, και προς όφελος της ε, πνευματικής μας ε, ηγεσίας. Τι θέλω να πω, θέλω να πω να έχετε και να επεξεργαστείτε ειδικά προγράμματα για τα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα. Ένα λεπτό παρακαλώ να είναι οι ερωτήσεις γιατί αν μιλάτε παραπάνω δεν θα έχει χρόνο η ε, υπουργό να απαντήσει. Σλοβενία. Ο κ. Σβέν, πρώην υπουργό Παιδείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Υπουργό για το ότι ε, παρουσίασε πολύ καλά τις προτεραιότητες του προγράμματος της, κυρίως ε, η μεταρρύθμιση Μπολόνια. Είναι πολύ σωστή. Τα πανεπιστήμια πρέπει να ανοίξουν για την αγορά και για την οικονομία. Το κράτος εμπλέκεται πάρα πολύ στο χώρο των πανεπιστημίων. Το κράτος ε, πρέπει να φύγει από αυτό το χώρο. Άλλοι τρόποι και κονδύλια χρηματοδότησης πρέπει να ζητηθούν, όχι από το κράτος και μόνο έτσι τα ε, πανεπιστήμια θα, είναι, ε, θα έχουν αυτοδιάθεση και θα είναι ανεξάρτητα από το κράτος. Πρέπει να προσεγγίσουμε τη δυτική μορφή πανεπιστημίων και μόνο με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη θα έχει πανεπιστήμια που θα κατατάσσονται ανάμεσα στα πρώτα δέκα του κόσμου. Παλιά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Humboldt, παραδείγματος χάρη, εξακολουθεί να υπάρχει ε, στο πανεπιστήμιο αυτό ε, ναι μεν εμπλέκεται το ε, κράτος αλλά επιτρέπει μία κατά το μάλλον ήτον αυτοδιάθεση των καθηγητών και των φοιτητών. Μόνο με την ε, εξέλιξη που σας είπα στον χώρο των πανεπιστημίων θα καταστεί δυνατόν να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην Ευρώπη ανάμεσα στην ε, παραγωγή και στα προϊόντα που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ο κύριος Μπίσκι από τη Γερμανία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που μας είπατε ε, και έχω όμως κι εγώ μία παράκληση. Σλούμπιτσε. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα που δείχνει ε, ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε και της βιατρίνα, γιατί η βιατρίνα ε, βοηθάει την ανταλλαγή την πολιτιστική. Πολύ καλή αυτή η βιατρίνα και για την Πολωνία και για τη Γερμανία. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε τη βιατρίνα. Το δεύτερο που θέλω να πω ε, έχει σχέση με την τέχνη. η πρόεδρος διακόπτη, ε, ο κ. Μπίσκι. Κοιτάξτε, η Πολωνία έχει καταπληκτική εκπαίδευση στον τομέα του κινηματογράφου και της μουσικής. Γι' αυτό λοιπόν ε, σκεφτείτε ότι η Πολωνία έχει να προσφέρει κάτι στην Ευρώπη πολύ περισσότερο από άλλα κράτη. Άλλα κράτη δεν διαθέτουν αυτές ε, τις ε, δυνατότητες της Πολωνίας. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ χαιρετίζω την παρουσία εδώ των εκπροσώπων της Πολωνικής Προεδρίας στην οποία εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχω κάποια αμφιβολία ως προς το κατά πόσον πρέπει να δοθεί τόση σημασία στο πρόγραμμα Έρασμος για τις γειτονικές μας χώρες. Νομίζω ότι το δυναμικό του έχει φτάσει στα όρια του. Ίσως να μην το εννοούσε όπως εγώ η πρόσωπος της Προεδρίας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τις ανταλλαγές φοιτητών μέσα στην Ένωση. Έπειτα, οι δικαστές και οι ανθρακορίχοι είναι επαγγέλματα που και αυτά χρήζουν μεταρρύθμισης. Μπορεί να είναι κάτι πολύ δύσκολο αλλά απαραίτητο. Και αφού ζητάμε αμοιβαία αναγνώριση προσόντων πρέπει να δούμε την πραγματική ζωή και την πραγματική κατάσταση χωρίς να κλεινόμαστε σε αφηρημένες ιδέες. Έπειτα, το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να έχει και αυτό σχέση με την πραγματικότητα και τρίτον, ο χρόνος διδασκαλίας είναι επίσης κάτι σημαντικό. Μερικοί καθηγητές διδάσκουν πολύ λίγο, τα αφήνουν όλα στους φοιτητές να κάνουν μόνοι τους την έρευνά τους. Ακόμη και για τους μαθητές στα δημοτικά επειδή είναι πολύ λίγοι οι δάσκαλοι αναγκάζονται να αφιερώνουν πάρα πολύ λίγο χρόνο στην πραγματική διδασκαλία. Μόνο αν έχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι τον απαραίτητο χρόνο για να διδάξουν θα μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε τα σχολεία όπως πρέπει. E, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ την ε, Υπουργό για την ε, παρουσίασή της ε, ιδιαίτερα διότι μίλησε για τις, ε, ε, τη γνώμη της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και πόσο σημαντική είναι για το, αυτή η γνώμη για το Συμβούλιο. Ήσασταν Ευρωβουλευτής για τρία χρόνια πριν γίνεται υπουργό, το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω ότι θα επηρεάσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ για τη δήλωση επίσης ότι θέλετε να προστατεύσετε προγράμματα όπως το Erasmus και το Comenius. Ελπίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση θα αποτελέσει μήνυμα προς την Πολωνική Προεδρία. Το περιεχόμενο είναι σημαντικό, αλλά και το όνομα είναι σημαντικό. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ασφαλώς είναι πολύ δύσκολη η μεταρρύθμιση τη ανώτατης εκπαίδευση. Θα Πρέπει να δώσουμε όμως σημασία σε αυτό που ο κύριος Φίσας εξέλα, Στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις και με την οικονομία γενικότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης της αυτονομίας των κρατών μελών. Και βέβαια θέλουμε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να είναι ανταγωνιστικά όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Γνωρίζετε τον κατάλογο «Τσανγκάι» το κατάλογο τη ε, εκεί θα πρέπει τα πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό τομέα τη πολιτική στην Ευρώπη. Νομίζω όμω ότι του φιλόδοξου στόχου του 2020, κυρίω όσον αφορά τη μείωση τη ανεργία των νέων στην Ευρώπη, του στόχου αυτού, δεν θα μπορέσουμε να του πετύχουμε εάν δεν ασχοληθούμε και με την επαγγελματική κατάρτιση. Γι' αυτό λοιπόν θα σα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων αν μπορούσατε να αναφερθείτε στην επαγγελματική κατάρτιση, ε, κυρίω στο πρόγραμμα Leonardo da Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα έτσι ώστε η να προσφέρεται όχι μόνο στους ε, φοιτητές πανεπιστημίων αλλά και σε νέους ανθρώπους ε, που βρίσκονται στον χώρο της επαγγελματικής ε, κατάρτισης. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα ή που δημιουργείται πρόβλημα είναι εκεί όπου αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε από την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να συντονίζονται καλύτερα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε τα πρακτικά προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή του προγράμματος Λεωνάρντο να τα λύσουμε οι δυνατόν έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι ακόμα πιο επιτυχημένο από ό,τι ήδη είναι. Πρόεδρος, ε, βέβαια αυτό δεν είναι δουλειά ε, της Υπουργού. Ε, αυτή είναι μια ερώτηση περισσότερο προς την κυρία Χαλ. Τώρα είναι πολύ αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει βέβαια τους συνεργάτες της θα τα σημειώσουν ε, φαντάζομαι. Βλέπω τα πρόσωπά τους, εκπέμπουν ε, επιτυχία και νομίζω θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Τάκουλα έχει το λόγο. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό για όλα αυτά που μας είπε και πρέπει να πω έχοντας ε, κατά νου τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια νομίζω ότι τα πανεπιστήμια αυτά πρέπει ε, να παρουσιάζουν ε, ενδιαφέρον ε, και για φοιτητέ από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία, γιατί όχι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα αποτελούσε λόγο τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη να γίνουν πιο ενδιαφέροντα εάν πραγματικά επιθυμούμε να ελοποιήσουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας, δηλαδή αν θέλουμε να γίνουμε μια κοινωνία που να βασίζεται στη γνώση, τότε χρειαζόμαστε τα πανεπιστήμια και χρειαζόμαστε καλά πανεπιστήμια. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να πω ότι σημαντικότερο από το όνομα και το σήμα είναι το περιεχόμενο. Αυτό, σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε υπό την Πολωνική Προεδρία έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε νέο περιεχόμενο στα προγράμματα. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Όχι απαραίτητα να κολλάμε στα ονόματα και στα σήματα. Η κυρία Χαλ ε, αναφέρθηκε ήδη στο θέμα αυτό. Ας πάμε στο πρόγραμμα Comenius. Εκεί μπορούμε να προσθέσουμε αξία. Μπορούμε ε, να εξελίξουμε περαιτέρω την όλη διαδικασία. Παραδείγματο χάρη η εκμάθηση γλωσσών. Ένα παιδί στην Πολωνία, στην τέταρτη τάξη, αν θέλει να προχωρήσει, ε, χρειάζεται νέα ερεθίσματα. Άρα δηλαδή πρέπει να προσφέρουμε νέο περιεχόμενο στα προγράμματα. Ε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να μην παραμένουμε ε, προσδεδεμένοι στα παλιά ονόματα. Σε ένα λεπτό βέβαια δεν μπορώ να πω όλα αυτά που σκέφτομαι, αλλά ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της ε, Πολωνικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για το περιεχόμενο. Η κυρία Βεναλόβα. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Αφού μιλάμε για εξέλιξη του Εράσμου, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης του προγράμματος. Ελπίζω υπό την Προεδρία σας να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, <coughs> αλλά η έλλειψη πόρων Πιστεύουμε ότι αν θέλουμε περισσότεροι φοιτητέ να ασχοληθούν με το πρόγραμμα έρασμο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν, να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους σε αυτό. Αφού μιλάμε δε για την εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων μεταξύ φοιτητών από διαφορετικές χώρες αλλά και στην ίδια χώρα. Μάλιστα, κυρία Υπουργέ μου. Ευχαριστώ πολύ για όλα σας τα ερωτήματα. Μερικά ήταν παραπλήσια, θα τα απαντήσω μαζί λοιπόν. Για τον έρασμο και την κινητικότητα, ο κύριος Κέλλη και η κυρία Νεβεντάλοβα είπαν ότι πιο σημαντικό είναι να ενδυναμωθεί, να διευρυνθεί το έρασμος μέσα στην Ένωση και να μην τονίζουμε τόσο πολύ την πολιτική γειτονία. Η κυρία Νεβεντάλοβα μάλιστα είπε ότι χρειάζεται και περισσότερη εσωτερική χρηματοδότηση για τη διεύρυνσή του εσωτερικά. Συμφωνώ βέβαια. Συμφωνώ και πάνω απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί το πρόγραμμα Έρασμος εσωτερικά. Το, το δέχομαι αυτό. Να μην απευθύνεται πλέον μάλιστα μόνο σε φοιτητέ που σπουδάζουν για το πρώτο τους δίπλωμα αλλά και, για και σε μεταπτυχιακούς για μάστερ και διδακτορικό. Άλλο στοιχείο, η διεύρυνσή του προς τις χώρες γειτονίας. Δεν εννοούσα ότι το πρόβλημα είναι η διαρροή, η ροή εγκεφάλων. Ορισμένες χώρες της Ένωσης που έχουν κάπως πιο αδύνατα πανεπιστήμια μπορεί να καταλήξουν με διαρροή εγκεφάλων και εσωτερικά πρέπει κανείς να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει σε χώρα διαφορετική από τη δική του. Και η διαδικασία της Μπολόνιας προέβλεπε τουλάχιστον 20% των φοιτητών να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Γιατί έτσι διευρύνουν τους πνευματικούς των ορίζοντες. Αποκτούν νέα προσόντα, νέο είδος γνώσης, περισσότερη γνώση. Αυτό το επεξεργαζόμαστε. Καλό θα ήταν το κοινοβου... και τα κοινοβούλια, οι βουλές, να το σκεφτούν. Είναι ένα από τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του προγράμματος Έρασμος. Τι ποσοστό δηλαδή φοιτητών εποφελούνται για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Άλλο. Μιλήσατε για κάτι πολύ επώδυνο για όλους μας, ιδιαίτερα για τις καινούργιες χώρες μέλη. Πολλοί αποφυτούν πηγαίνουν σε κάποια γειτονική χώρα και διαπιστώνουν ότι αναγκάζονται να γίνουν ταξιτζίδες. Το είπε και η πρόεδρος. Και εμείς στην Πολωνία το λέμε ότι αναγκάζονται πολύ μορφωμένοι να πλένουν πιάτα σε εστιατόρια. Το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων λοιπόν είναι ένα από τα θέματα κλειδιά για την Ένωση και την Κομισιόν της. Ξέρω ότι το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων θα είναι από τα κυριότερα θέματα που θα προτείνει η Κομισιόν τον Δεκέμβριο. Προς το παρόν όμως οι χώρες μέλη, οι χώρες μέλη ήδη επεξεργάζονται ένα πλαίσιο διευθέτησης των προσόντων στην Ευρώπη για να επιτρέπεται όχι μόνο η αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων ενός χαρτιού δηλαδή μιας περγαμηνής αλλά και αναγνώριση εμπειρίας όταν έχει μάθει κανείς κάτι κάπου να αναγνωρίζεται η μάθηση αυτή και αλλού ας πούμε κάποιος που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ στη Γερμανία να αναγνωρίζονται τα προσόντα του όπως και του πτυχιούχου από ένα μικρό πανεπιστήμιο της Πολωνίας μπορεί να μην είναι της ίδιας ποιότητας τα πανεπιστήμια αλλά να αναγνωρίζονται εσπουδέ. Κυρία Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχουμε, πόσο χρόνο έχουμε. Α, τότε καλά. Μπορώ να απαντήσω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Τότε. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο αυτό το κοινό πλαίσιο αναγνώρισης προσόντων είναι τόσο σημαντικό. Γνωρίζουμε τη διαδικασία της Μπολόνια, γνωρίζουμε και τις ελλείψεις της που οφείλονται στην πολλαπλότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων στις διάφορες χώρες ή μεταξύ των διαφόρων χωρών. Δεν πρόκειται βέβαια να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα για ολόκληρη την Ένωση, δεν γίνεται αυτό. Αλλά επειδή η Πολωνία προεδρεύει και της διαδικασίας της Βολωνίας θα προσπαθήσουμε να μεταρρυθμίσουμε αυτά που αποφασίστηκαν εκεί για να δημιουργηθεί τουλάχιστον η δυνατότητα πιο εύκολης αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται καλύτερη κατανομή μεταξύ των πανεπιστημίων σε ανακατηγορίες επαγγελματικά, επαγγελματικές σχολές, τεχνικές σχολές, ανώτατα ιδρύματα κτλ. Και έρχομαι τώρα στο ερώτημα του κυρίου Βίσκη. Ε, Για το Πανεπιστήμιο Βιαντρίνα. Η χρηματοδότηση από δύο γειτονικέ χώρες είναι κάτι το πολύ ωραίο. Η Βιαντρίνα e, μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας από κοινού ενέκριναν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καταπληκτικό δηλαδή παράδειγμα τέτοιας κοινή πρωτοβουλία και θα έπρεπε να πολλαπλασιαστεί και αλλού γιατί εδώ συνδυάζονται κρατικά κονδύλια και άλλα κονδύλια. Είναι λοιπόν σημαντικό τα διαρθρωτικά κονδύλια, κρατικά και ενωσιακά, να μπορούν όπως στην Πολωνία, Πολωνία να χρησιμοποιούνται για να, για να μειωθεί η ανεργία των διπλωματούχων και πτυχιούχων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνο όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό αλλά και στη δική τους χώρα. Η χρησιμοποίηση λοιπόν των διαρθρωτικών ταμείων έτσι ώστε να γίνονται επενδύσεις στα τεχνικά, στις τεχνικές σχολές και πανεπιστήμια θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους φοιτητές και φοιτήτριες να σπουδάζουν στους τομείς όπου θα μπορούν να βρουν δουλειά. Dużo więcej Στην Πολωνία μετά από ένα και μόνο χρόνο αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητών στα τεχνικά πανεπιστήμια περισσότερο από ότι σε παιδαγωγικά θέματα, θεωρητικά θέματα όπου δεν υπάρχει δουλειά. Περισσότεροι φοιτητέ και φοιτήτριε λοιπόν στα τεχνικά πανεπιστήμια. Ξέρω ότι δεν απάντησα σε όλα σας τα ερωτήματα γιατί υπήρχαν και μερικά για την προσαρμογή στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Το πρόγραμμα Μαρία Κιουρί, ας πούμε, είναι κάτι που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και σε αυτό. Γιατί και η Μαρία Κιουρί ήταν Πολωνή. Γι' αυτό του δίνουμε σημασία. Και θέλουμε να οργανωθεί μια συνάντηση, μια, ένα συνέδριο όσων ασχολούνται με το πρόγραμμα αυτό στη Βαρσοβία γιατί ελπίζουμε να συνεχιστούν τέτοια προγράμματα που τονίζουν, που αφορούν βέβαια ιδιαίτερα την έρευνα. Και κάτι ακόμα, κάτι ακόμα. Το σημαντικό με τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα, τα ανώτατα ιδρύματα, είναι το περιεχόμενο των σπουδών. ξεχνάμε συνήθως ότι υπάρχει και το θέμα της μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Στο σημερινό κόσμο με τις νέες του τεχνολογίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και αυτό μια πρόκληση για μας. Τέλος, τέλος. Μίλησα για ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. φαίνεται ότι e, προτάσεις όπως τη διάσκεψη που θα οργανωθεί στην Κρακοβία είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα ως προς το πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών στην Ένωση για την έρευνα ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στην Προεδρία μας. Ευχαριστώ πολύ και μία τελευταία φράση. Έχω συνεννοηθεί, ήμουν και εγώ κάποτε βουλευτής και έθετα ερωτήματα σε υπουργούς όπως κάνετε σήμερα και εσείς και γι' αυτό ήταν τόσο ενδιαφέρον για μένα σήμερα η συνάντησή μας. Ελπίζω η δουλειά σας να είναι πάντοτε καρποφόρα για την Ευρώπη και τους πολίτες της ε, και ελπίζω η συνεργασία μας τους επόμενους έξι μήνες να είναι πολύ θετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα είναι πολύ δύσκολο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να εξετάσουμε όλα τα θέματα. Αλλά θέλω να δώσω μια απάντηση στον κύριο Κέλλη. Αγαπητέ Ζαν, το ε, θέμα του προγράμματος Εράσμους δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε εγωιστικά. Το πρόγραμμα Εράσμους είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν ε, συμμετέχουν ε, γειτονικές χώρες αυτές πρέπει να πληρώσουν. Πληρώνουν βέβαια εν μέρη από τα προενταξιακά κονδύλια ας πούμε των Βαλκανίων και από κονδύλια που πηγαίνουν σε τρίτες χώρες. Δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα στον προπολογισμό μας, απλά ανοίγει ορίζοντας ο δικός μας και των άλλων. Ε, να μην σκεφτόμαστε, λοιπόν ε, τόσο κοντόφταλμα. Αν δεν μπορούμε να ε, εντάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα μέλη, τα κράτη της Ευρώπης, τουλάχιστον ας πούμε να έχουμε μια πολιτιστική ανταλλαγή. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε τώρα στον κύριο Τσουχόφσκι. Αναπληρωτής, ε, μάλλον αναπληρώνει υπουργό που είναι ε, άρρωστος. Δίνω το λόγο στον κύριο Τσουχόφσκι. το αφεντικό σας είναι ο κύριος Ντρογεύσκι, έτσι δεν είναι, ωραία. Έχετε το λόγο. E, Πράγματι, το άτομο το οποίο θα πρέπει να παρουσιάζει τι ε, προτεραιότητε τη Πολωνική Προεδρία ε, ε, στον τομέα τη εθνική κληρονομιά και του πολιτισμού είναι ο κ. Μπόγκταν Ντρογεύσκη, ο οποίο έπεσε θύμα ατυχήματο δυστυχώ. Ε, μας ακούει βέβαια μέσω ίντερνετ από το νοσοκομείο. Και στέλνει τους χαιρετισμούς του και τους στέλνουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας. Κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα τις προτεραιότητες της ε, Πολωνικής Προεδρίας στον τομέα του πολιτισμού και, της, ε, και των οπτικοακουστικών. Η βασική προτεραιότητα στον τομέα της, ε, του πολιτισμού είναι ο ρόλος του πολιτισμού στη δημιουργία διανοητικού κεφαλαίου στην Ευρώπη είναι κομμάτι των οριζόντιων, ε, της οριζόντιας ε, προτεραιότητας της ε, Πολωνικής Προεδρίας για την δημιουργία ε, διανοητικού κεφαλαίου και έχει σχέση με την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων όπως η συνειδητοποίηση του πολιτισμού, της κουλτούρας. Το διανοητικό κεφάλαιο είναι όλα, όλες οι άειλες ε, διανοητικές ικανότητες ε, που μπορούν να αποκτηθούν και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραμείνει καινοτόμα, αν θέλει να μπορεί να υλοποιεί στόχου όπως αυτού τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 100% του διανοητικού μας κεφαλαίου. Το διανοητικό μας κεφάλαιο αποτελεί κοινή μας επένδυση για το μέλλον πολιτιστικές ε, ικανότητες και δεξιότητες δίνουν στους πολίτες την δυνατότητα να σκέφτονται με ένα καινοτόμο τρόπο, να είναι καινοτόμοι, να είναι δημιουργικοί. Αυτό είναι χρήσιμο όχι μόνο στις τέχνες, αλλά και στην επαγγελματική ζωή και στην ε, επιχειρηματική ζωή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν αποδείξεις ότι ε, παιδιά τα οποία ακολουθούν παρακολουθούν μαθήματα θεάτρου ε, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κατανοούν καλύτερα την άποψη των άλλων και αναπτύσσουν επικοινωνιακές ικανότητες πολύ περισσότερο από ότι παιδιά που δεν παρακολουθούν μαθήματα θεάτρου. Τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν μαθήματα θεάτρου θα αντιληφθούν σύντομα στο μέλλον ότι οι πρόσθετες ικανότητες που αποκτούν, τους δίνουν προβάδισμα και στην επαγγελματική ζωή. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πρότεινε συμπεράσματα ε, τα οποία θα αναφέρονται σε συνέργεια ανάμεσα στην, ε, στον πολιτισμό και την ε, καινοτομία, την έρευνα, την επιστήμη αφετέρου. Θέλουμε να μειώσουμε επίσημα με αυτόν τον τρόπο ε, τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να αυξήσουμε την απασχολησιμότητα ε, των ε, πολιτών μας και να βελτιώσουμε τη θέση του πολιτισμού στην μη τεχνολογική καινοτομία και να εντάξουμε τον πολιτισμό στη νέα γενιά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, Ακόμα θυμόμαστε τη συζήτηση για την δημιουργία της, ε, του Ευρωπαϊκού Σήματος Πολιτικής Κληρονομιάς. Ε, για μας ε, θα είναι μια δράση προτεραιότητας. Χαιρόμαστε που κατά τη διάρκεια τη Ουγγρική Προεδρία, ε, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό για αυτή την πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω ε, να ευχαριστήσω την κυρία Παλιαδέλη ε, που ήταν η συγγήτρια και την κυρία Πακ την πρόεδρο. Το κείμενο εγκρίθηκε πολιτικά αλλά χρειάζεται να το επεξεργαστούμε περισσότερο για να καταλήξουμε στην οριστική απόφαση. Σε μερικές μέρες, στις 18 Ιουλίου συγκεκριμένα, το Συμβούλιο θα υιοθετήσει το προσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση και το Συμβούλιο θα το λάβει στις αρχές Σεπτεμβρίου μια γρήγορη υιοθέτηση του κειμένου στη δεύτερη ανάγνωση από το Κοινοβουλίο θα επιτρέψει στην απόφαση αυτή να αρχίσει να εφαρμόζεται στο τέλος του χρόνου. Εν τω μεταξύ, η Πολωνική Προεδρία θα ξεκινήσει συζητήσει στο Συμβούλιο για την διαδικασία ε, διορισμού εμπειρογνωμόνων που θα έχουν ως καθήκον την, ε, ε, μάλλον στο, πάνελ ε, των 15 μελών για την έγκριση αυτού του Ευρωπαϊκού Σήματος Πολιτικής Κληρονομιάς. τα κριτήρια επιλογής των μελών σύμφωνα με την απόφαση θα γίνουν πλήρως σεβαστά από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διορισμών. Κυρίες και κύριοι, η απουσία συγκρίσιμων βιώσιμων στατιστικών στον τομέα του πολιτισμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίσουμε ε, στο να αποδείξουμε ότι η πολιτική πολιτική πραγματικά λειτουργεί. Για να αποδείξουμε ότι λειτουργεί η πολιτιστική πολιτική για να αποδείξουμε ότι ο πολιτισμός βοηθάει στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 2020 χρειαζόμαστε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Χωρίς αυτού του είδους τις αποδείξεις πώ ε, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο πολιτισμός είναι κάτι σημαντικό. Είναι κενά λόγια. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι ισχυρισμοί τέτοιου τύπου χωρίς στατιστικά στοιχεία δεν γίνονται πιστευτοί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν επανειλημμένως έχουν ζητήσει ε, την χρήση τέτοιων ε, συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και των αντίστοιχων μεθοδολογιών. Η Eurostat ξεκίνησε ένα project για πολιτιστικά στατιστικά στοιχεία το 2009. Το πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα ε, υποβληθεί το Σεπτέμβριο στο, στην, σε μια διάσκεψη η οποία θα ε, ε, λάβει και τις τελικές αποφάσεις προκειμένου να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε Ε, θα προτείνουμε μάλιστα στους υπουργού πολιτισμού να συζητήσουν το θέμα των πολιτιστικών στατιστικών κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του Νοεμβρίου. Ε, επιθυμούμε να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θα τονίζει ότι χρειάζεται να επεξεργαστούμε περισσότερο το θέμα αυτό, την, ε, αυτή την πτυχή των δραστηριοτήτων μας. Κυρίε και κύριοι, συνεργασία με τις, η συνεργασία με τις χώρες της ανατολικής, ε, τις ανατολικές γειτονικές μας χώρες είναι προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Το πιο σημαντικό γεγονός, να σας παρουσιάσω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουμε προγραμματίσει κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Την περασμένη εβδομάδα στη Βαρσοβία έλαβε χώρα μια διάσκεψη για την ανατολική διάσταση της κινητικότητας. Ήδη ε, μια προηγούμενη ομιλήτρια το ανέφερε. Τέσσερα Υπουργεία διοργάνωσαν αυτή τη διάσκεψη σε συνεργασία με την Κομισιόν για να ενισχύσουμε την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της νεότητας και του αθλητισμού. Πρόκειται για μια συνεργασία με τις, ε, τους ανατολικούς μας γείτονες της χώρας του Καυκάσου. Ε, κάτι τέτοιο θα θα οδηγήσει, ανοίγει το δρόμο για ένα φόρουμ στο τέλος Σεπτεμβρίου ε, σε, όπου θα συμμετέχουν οι ανατολικές γειτονικές μας χώρες και θα συζητήσουν πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη ε, σχέση συνεργασίας. Ε, τέλος ε, Νοεμβρίου προετοιμάζουμε ένα άλλο φόρουμ ε, της κοινωνίας των πολιτών και ε, θα ληφθούν εκεί υπόψη όσα θα έχουν συζητηθεί όπως επίσης θα ληφθούν υπόψη και στο Συμβούλιο των Υπουργών το Δεκέμβριο. Ελπίζω ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες οι σχετικές με την ε, γειτονική σχέση με τις ανατολικές χώρες θα ενισχύσουν την συνεργασία με τις χώρες αυτές και θα διευκολύνουν την ε, υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις ε, ανατολικές γειτονικές μας χώρες. Τώρα, προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο σε σχέση με τον τομέα των οπτικοακουστικών. Η βασική προτεραιότητα θα είναι η ψηφιοποίηση και η προστασία της πολιτικής κληρονομιάς. Πιστεύουμε ότι η ψηφιοποίηση και η διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές είναι απόλυτη προτεραιότητα, πολύ σημαντικό για όλη την κοινωνία μας. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μας επιτρέπουν όχι μόνο ε, να αποθηκεύουμε βιβλία, ταινίες, εικόνες, μουσική, φωτογραφίες κλπ. Αλλά επιτρέπουν ταυτόχρονα στους Ευρωπαίους και στους πολίτες όλου του κόσμου να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε όλα αυτά τα έργα. Πρέπει βέβαια να αναπτύξουμε και τις ικανότητες των χρηστών ε, στον, ε, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η πρόσβαση είτε αφορά εμπορική είτε αφορά προσωπική χρήση. Μπαίνοντα στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε μπροστά μας ε, καινούριες προκλήσεις σε ό,τι αφορά το ρόλο των πολιτιστικών ε, θεσμών και ιδρυμάτων για την πρόσβαση στην πολιτική κληρονομιά. Γι' αυτό τον λόγο η Κομισιόν το 2010 δημιούργησε μια ομάδα σοφών που εργάζεται, ε, επεξεργάζεται προτάσεις για το θέμα της ψηφιοποίησης. Τον Ιανουάριο 2011 αυτή η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση με τον τίτλο «Νέα Αναγέννηση» Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις για την online ε, ψηφιοποίηση και πρόσβαση προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνική Προεδρία θα εργαστεί επίσης επί του project Europalia και της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Επίσης θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες επί μιας οδηγίας που αφορά τα ορφανά έργα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα, το, το, την πτυχοακουστική πτυχή της οδηγίας. Ε, η, αν λύσουμε το πρόβλημα της μεταφοράς των δικαιωμάτων, μεταβέ των δικαιωμάτων, τότε η ψηφιοποίηση και ιδιαίτερα η, το, η Ευρωπάλια θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Ε, θα ανοίξει στο ευρύ κοινό με αυτόν τον τρόπο. Η πολιτική Προεδρία θα προτείνει η ψηφιοποίηση και η προστασία της πολιτικής κληρονομιάς ιδιαίτερος της οπτικοακουστικής πολιτικής κληρονομιάς ε, της κινηματογραφικής κληρονομιάς να συζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια μιας, άτι, ενός, μιας άτυπης συνάντησης που θα λάβει η χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου στο ε, Μπρέσλαου. Ε, η χρήση των ψηφιακών αρχείων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας θα συζητηθεί και ε, από εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός Ιουλίου. Ε, θα υποβάλουμε συμπεράσματα επίσης για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. θα προτείνουμε τέτοιου συμπεράσματα στο, στους υπουργούς. δύο συστήματα τάσει ε, είχαν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το, ε, το 1998 και το 2006. Αυτές οι συστάσει είχαν ως στόχο τη βελτίωση του επίπεδου προστασία των παιδιών και των νέων ε, στο ψηφιακό περιβάλλον. Η ψηφιακή εποχή έφερε αλλαγές στο οπτικοακουστικό περιβάλλον. Τα παιδιά έχουν πλέον εύκολη πρόσβαση σε προχωρημένες τεχνολογίες από μικρές ηλικίε. Πρόσβαση στο ίντερνετ όπου παίζουν παιχνίδια online, ακούν μουσική, αναζητούν πληροφορίες για τα project που τους έχουν αναθέσει στο σχολείο κλπ. Και επικοινωνούν με τους φίλους τους η κοινωνική δικτύωση ε, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ πλέον. 40% ε, περίπου των παιδιών σε ηλικίες 9 12 ε, και τα 2 τρίτα των παιδιών από, σε ηλικίες 12 με 16 έχουν προφίλ σε τέτοιου είδους δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η τηλεοράσεις ανταγωνίζονται με, τα, ε, με το ίντερνετ ε, προσφέροντας υπηρεσίες ε, pay-per-view on demand κλπ. Τα παιδιά όμως ενδεχομένως δεν γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους που συνοδεύουν τέτοιου είδους υπηρεσίες μέσω ίντερνετ ή μέσω τηλεόρασης. Γι' αυτό το λόγο ο γονικός έλεγχος, η, τα φίλτρα και άλλα μέσα προστασίας των ανηλίκων ε, είναι μερικά από τα μέτρα, μερικές από τις δραστηριότητες που θα προωθήσει η Πολωνική Προεδρία ανεξαρτήτως μέσου για να εξασφαλίσουμε υψηλό βαθμό προστασίας των παιδιών και των νέων. Κυρίες και κύριοι. Όπως ε, είπε, ε, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, ε, θέλουμε να δώσουμε σημασία στα προγράμματα Media, Media Mundus και Culture που είναι τα βασικά μας εργαλεία για την χρηματοδότηση του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιορτάζουμε την 20η επέτειο της ε, δημιουργίας του προγράμματος ε, Media που συνεισέφερε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ε, είναι ανυπολόγιστη η, ε, συνεισφορά του Media. Το ίδιο και για, την, και για το πρόγραμμα Culture που έχει υποστηρίξει πολιτιστικού φορείς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο τομεί αυτοί έχουν πλέον τα δικά, το δικό τους χρηματο, χρηματοδοτικό μέσο. Συνεπώς, ε, και οι δύο αυτοί ε, τομείς έχουν αποκτήσει ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το media και το culture και το Media Mundus θα λήξουν το 2013 όμως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα προγράμματα θα επηρεαστούν βέβαια από τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές για τα έτη 2014-2020. Η Πολωνική Προεδρία είναι πεπισμένη ότι οι πολιτικές δραστηριότητες και οι οπτικοακουστικές δραστηριότητες βρίσκονται στο κέντρο του ε, ευρωπαϊκού οράματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν να υποστηρίξουμε ε, τον πολιτισμό και τα μέσα με εργαλεία που θα δίδουν συνέχεια στα προγράμματα culture και media με επαρκή χρηματοδότηση στο, στο ε, κατάλληλο επίπεδο. Κλείνοντα, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για τη σκληρή δουλειά της, για τη συνέπειά της, για την αποφασιστικότητά της. Ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί πιο κατάλληλη στον πολιτισμό μέσα στην ατζέντα Ευρώπη 2020. Ε, επίσης για τις προσπάθειές τους ε, θα ήθελα να βοηθήσω τη Δανία και την Κύπρο για την συνεργασία τους ε, στη, στο πλαίσιο της, ε, του τρίο του των προεδριών. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένω την υποστήριξή σας, τη συνεργασία σας και βέβαια σας ε, καλούμε να μας επισκεφθείτε στην Πολωνία, να συμμετάσχετε στα πολιτικά ε, γεγονότα τα οποία στις πολιτικές εκδηλώσεις που οργανώνουμε. Ιδιαίτερως θα ήθελα να σας, ε, να σας καλέσω στον Πρέσλαο στον 8 με 11 Σεπτεμβρίου 2011. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Κύριε Υφυπουργέ, διορθώνει Πρόεδρος. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Καβαντά από τη Γαλλία. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που μια τόσο πολιτικά πλούσια χώρα όπως η Πολωνία ε, παίρνει την προεδρία ε, και θα προεδρεύσει και στο Συμβούλιο Πολιτισμού. Θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Οι νομοθετικές προτάσεις τάσεις για, το για τα πολιετή προγράμματα Culture και Media που θα, που θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί πέρσι από το Κοινοβούλιο. Θα μας ε, αποσταλούν το φθινόπωρο τελικά ή όχι. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι το πολιετές πρόγραμμα λύγει το 2013. Χρειάζεται από την άλλη μεριά και χρόνος για την προετοιμασία της τελικής έκθεσης. Συνεπώς, θα μπορούσατε να μας πείτε αν σήμερα Έχετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε το, το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και τρίτον πώς θα σας φαινόταν η ιδέα το media να συμπεριληφθεί στο culture με ένα καινούριο τίτλο culture media αντί να έχουμε ξεχωριστό πρόγραμμα media τρεις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις ευχαριστώ Madame Nevenalova, Επόμενη μιλήτρια από τη Σλοβακία. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ευχόμαστε στον Υπουργό σας ε, περαστικά. Καλή ανάρρωση. Ε, μου αρέσει πολύ το, το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας σας. Έχετε πολύ φιλόδοξους στόχους και ελπίζω να τους επιτύχετε. Και ελπίζω να δώσετε το καλό παράδειγμα. Γιατί πολύ συχνά σε περίοδους κρίσης γίνονται περικοπές. Εσείς μιλήσατε για το Ευρωπαίανα, για την ψηφιακή βιβλιοθήκη, τουλάχιστον αυτό ελπίζω να εννοούσατε. Και θα ήθελα να γνωρίζετε ποιοι να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι σας όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Ποια είναι τα σχέδιά σας, τα σχέδια υλοποίησης. Ακούσατε ότι η δική μας Επιτροπή ε, τάσεται υπέρ ε, του ε, βραβείου Λουξ. Αλλά ακούσαμε ότι μερικοί επιθυμούν να καταργηθεί το βραβείο αυτό και ελπίζω να μας στηρίξετε να μην καταργηθεί η Πρόεδρος. Το βραβείο Λουξ είναι δικό μας παιδί και δεν έχει καμία σχέση με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν. Η δικό μας είναι και μια χαρά είναι. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος των ε, φιλελευθέρων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για όλα αυτά που μας είπε γιατί επέδειξε ε, εμπειρογνωμοσύνη. Έχω να θίξω δύο θέματα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι το ατού της Ευρώπης ε, είναι ότι έχουμε μεγάλη πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Υπάρχει το, ε, η πολιτιστική κληρονομιά της ε, UNESCO, έχουμε ε, τη δική μας τη σφραγίδα πολιτιστικής λουμιάς. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, προσπάθειες. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες έτσι ώστε για την Ευρώπη να προκύπτει προστιθέμενη αξία. Μερικές φορές ε, έχουμε την αίσθηση ότι όσον αφορά αυτά τα προγράμματα μεγαλύτερος είναι ο ενθουσιασμός ε, από την τελική επιτυχία. Βεβαίως ε, και είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, για τον τουρισμό. Πάω τώρα στο θέμα της ψηφιακής κοινή αγοράς. Αυτός είναι βέβαια ένας σημαντικός τομέας και νομίζω ότι στον τομέα αυτό πρέπει να αναζητήσουμε νέα μέσα έτσι ώστε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ε, να είναι η αιχμή του δόρατος ε, στην ε, ψηφιακή κοινή αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία όθηση έτσι ώστε η ψηφιακή τεχνολογία και ο ψηφιακός πολιτισμός να μπορούν να διοδοθούν και πέρα από τα σύνορα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή την ψηφιακή κοινή αγορά πραγματικά να την οθήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ για το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα ως προς τον πολιτισμό. Και θα ήθελα να πω και εγώ προς τον κύριο Συντρογεύσκη που συνεργάζεται μαζί σας σε αυτό το πρόγραμμα να του μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μου. Το Σεπτέμβριο η Επιτροπή μας θα πάει στο Βρότσλαου και θα συζητήσουμε εκεί με διανοούμενους και διανοούμενες το ρόλο του πολιτισμού Άρα θα συνεχίσουμε κάπως τη σημερινή μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάντως και σας ενθαρρύνω κύριε Υπουργέ μου να σκεφτείτε το θέμα της παιδείας και του πολιτισμού. Το Την οπτικοακουστική πτυχή, τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο γιατί και εγώ είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε μια έκθεση που σε λίγο θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, όλα τα πολιτιστικά, οι δυνατότητες που πρέπει να έχει και να μπορεί να εκφράσει ο κάθε Ευρωπαίος και Ευρωπαία. Αυτό είναι σημαντικό για όλες τις χώρες γιατί εκτός από τη Γαλλία δεν υπάρχει πουθενά ε, εκπαίδευση ή παιδεία για τον πολιτισμό ειδικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το θίξατε και θέλω να σας ε, κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συνδέσατε τα πολιτιστικά προγράμματα με το πρόγραμμα Μίδια ώστε να υπάρχει καλύτερη στόχευσή τους. Δεν υπάρχει βέβαια είπατε επανάσταση, υπάρχει εξέλιξη, αλλά τα προγράμματα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα ιδίως στην οπτικοακουστική πλευρά τους. Και εμείς ως συνομοθέτες στην Ένωση ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα και αν σκεφτούμε τη δημιουργικότητα των Ευρωπαίων θα ήθελα να είστε και εσείς ιδιαίτερα άτεγκτος με τους υπόλοιπους υπουργούς για να επιμείνετε να χορηγηθεί η χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κέλλης. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό καταρχήν για την πολύ ωραία του παρουσίαση για τον πολιτιστική κληρονομιά, τα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Από την αρχή, στην αρχή μίλησε για στατιστικά στοιχεία ως προς την αξία των μαθημάτων, των θεατρικών μαθημάτων όπου υπάρχουν βέβαια. Θα ήθελα να ξέρω όμως πόσα τέτοια μαθήματα υπάρχουν στα γυμνάσια και τέτοιου είδους πολιτιστικές δραστηριότητες. Κάτι άλλο επίσης μίλησε για τη δημιουργία μιας ομάδας σοφών. Μήπως θα υπάρχει και καμία σοφή μεταξύ των σοφών αυτών. Μικρόφωνο παρακαλώ η Πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω θερμά τον Υπουργό. Έχω μία πολύ σύντομη ερώτηση. Εσείς ε, δυστυχώς ε, δεν μιλήσατε για τον οίκο της ε, ευρωπαϊκής ιστορίας. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Συμβουλίο ούτε με την Κομισιόν. Αυτό είναι δικό μας θέμα του Κοινοβουλίου. Διακόπτη Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ όμως θα ήθελα να ακούσω την άποψη του Υπουργού. Αυτό ήθελα. Κύριε Υπουργό, έχει το λόγο. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι όσον αφορά τον συνδυασμό προγραμμάτων. Ε, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που ελέγξαν και εγώ ίδιος έχω μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι έχουμε όλη την ίδια άποψη, έχουμε κατά νου προγράμματα ε, που λειτουργούν πολύ καλά στον τομέα του πολιτισμού όπως το πρόγραμμα Media ή το πρόγραμμα Media Mundus ε, τα προγράμματα αυτά πράγματι ε, είναι αναγνωρίσιμα και είναι σημαντικό να διατηρήσουμε προγράμματα τα οποία λειτουργούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Όταν ε, ένας ε, παραγωγός αποφασίζει να γυρίσει, να χρηματοδοτήσει μία ταινία, όλα αυτά τα προγράμματα παίζουν σημαντικό ρόλο. Ε, και αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά είναι να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Ε, το να επιχειρήσουμε κάτι καινούριο, αυτό πάντα ενέχει κινδύνους. Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά μπορώ να σας πω ότι εγώ ε, συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικά, ότι Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι γνωστά, αναγνωρίσιμα σήματα που λειτουργούν σωστά και δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα. Γιατί πολύ συχνά το τέλειο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ο εχθρός του καλού. Στην επόμενη ερώτηση που ετέθη σχετικά Τικά με την Ευρωπαϊκή. Υπήρξε κάποια στιγμή όπου η Ευρώπη ε, ασχολήθηκε σε βάθος ε, με το πρόγραμμα αυτό. Ε, εγώ όμως ως υπουργό Πολιτισμού έχω να αντιμετωπίσω και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν πρόκειται λοιπόν για συνδυασμό βιβλιοθηκών και αρχείων, εκεί ανακύπτει το πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αν λοιπόν επιθυμούμε να εφαρμόσουμε σωστά το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά, πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος, έτσι ώστε το πρόγραμμα να εφαρμόζεται ικανοποιητικά. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εφαρμόσουμε την οδηγία εκείνη που αφορά πολλά προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό, όπου δηλαδή ε, πρόκειται για ε, το να καταστούν πιο προστά έργα που έχουν σχέση με την ε, ψηφιοποίηση. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη. Και ο κύριος Τακούλα τοποθετήθηκε επί του θέματος. Και εγώ λοιπόν ε, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Πακ. Και κάτι άλλο. Ε, η σφραγίδα ευρωπαϊκής ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό το σήμα έχει σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ε, έχει, υπάρχει βέβαια και ε, η σφραγίδα ποιότητα τη UNESCO, είναι όμως σημαντικό να έχουμε και τη δική μας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία και αυτό που ενδιαφέρει είναι τι επιδιώκουμε. Αν επιδιώκουμε μια, ένα σήμα ποιότητας της ευρωπαϊκής ε, πολιτιστικής κληρονομιάς, τότε πρέπει να αναθέσουμε σε εμπειρογνώμονες, σε ειδικού να βρουν έναν τρόπο να προβάλλουν αυτή την ιδέα της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Και τη σφραγίδα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα την πάρουν μόνο τα καλύτερα προγράμματα. Άρα δηλαδή οφείλουμε να βρούμε μια καλή ιδέα για το ποια προγράμματα πρέπει να λάβουν αυτή την σφραγίδα ποιότητας. Βεβαίως ε, είναι σημαντική και το γεωγραφικό στοιχείο, η γεωγραφική διάσταση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ε, ποιότητα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και κάτι άλλο. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να θίξουμε. Αφενός έχουμε τον μύθο αυτό της Ευρώπης σχετικά με την ίδρυση Ευρώπης που είναι άρρηκτα συνδεμένος με την ελευθερία. Από την άλλη όμως, και βλέπουμε ότι αυτό έχει άμεση σχέση με την ψηφιακή εποχή, από την άλλη λοιπόν διαπιστώνουμε ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια ε, παράδοση η οποία προβλέπει και την προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Ο δημιουργός ε, πρέπει να είναι ο μόνος ιδιοκτήτης ε, δικαιωμάτων στο έργο του. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στα, στα έργα τέχνης η μόνη δυνατότητα είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Και αυτό είναι προς όφελος των δημιουργών. Πρέπει να τους επιτρέπουμε την όσο καλύτερη πρόσβαση στα έργα τους. Υπάρχουν κάποιες σχετικές απόψεις που έχουν εκφραστεί επί του θέματος, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος. Εγώ σας ε, επαναλαμβάνω, η δική μας προτεραιότητα και η δική μας άποψη είναι ότι ο δημιουργός είναι ο ένας και μόνος ε, ιδιοκτήτης ε, των πνευματικών του δικαιωμάτων. Επίσης αναφέρθηκα και στην προστασία νέων και ενηλίκων στο διαδίκτυο, που είναι χρήστες του διαδικτύου. Πρέπει να έχουμε έναν κατάλογο ε, ασφαλών ε, έργων. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να παρεμβαίνουμε στην ελευθερία των πολιτών. Ο κύριος ε, Μπόρις, κύριε Μπόρις, και εσείς κάνατε κάποιες παρατηρήσεις. Πράγματι, αν σκεφτεί κανείς τα διάφορα προγράμματα, είναι σημαντικό οι αλλαγές να γίνουν σταδιακά και όχι καταιγιστικά. Και μου τέθηκε άλλη μια ερώτηση που αφορά στα στατιστικά δεδομένα. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ζητήσω τη βοήθεια της συνεργάτητος. Ε, υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν γίνει και στην Πολωνία ετέθη ένα ερώτημα σχετικά με την εκπαίδευση ε, για θέματα πολιτισμού. Αυτό όμως είναι αρμοδιότητα σχολείου. Εμείς έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα Όλα αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες ε, του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό σχολικό σύστημα όπως σας είπα και κατόπιν τούτου εμείς στην Πολωνία είμαστε σε θέση να εκπαιδεύουμε ε, θαυμάσιους μουσικούς. Στον Μπόζαρ ε, θα δείτε μία θαυμάσια έκθεση Πολωνών καλλιτεχνών. Όλοι αυτοί είναι απόφοιτοι της ε, δικής μας της σχολής καλών τεχνών. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πραγματικά ε, και ουσιαστικά αναφέρομαι στην ε, εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού. Κατόπιν του κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά την τέχνη που μας προσφέρει η Πολωνία ε, και σας συστήνω ε, να πάτε σε αυτή την έκθεση στο Πόζα. Ε, σήμερα το βράδυ θα γίνουν και τα γένεια μιας έκθεσης. Εγώ θα πάω και καλό και τους άλλους γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι γιατί ετέθη το θέμα. Όσον αφορά το πρόγραμμα Media, το γεγονός ότι έγκαιρα ε, σημάναμε συναγερμό οδήγησε ώστε το πρόγραμμα αυτό δεν θα εξαφανιστεί, θα υπάρξει τέτοιο πρόγραμμα. Ε, γι' αυτό το λόγο είχα ε, χτε μια συζήτηση με την Κομισιόν. Άρα δηλαδή μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Καταρχήν θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Κατά δεύτερον, σε αυτό το πακέτο διασφαλίζεται το πρόγραμμα Media. Άρα δηλαδή Ξέρουμε πολύ, πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα Media και σε σχέση με το βραβείο Lux. Δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε άλλο. Χθε είπα στον αρμόδιο ότι δεν είναι δυνατόν να έρθετε το ε, Νοέμβριο και να μας υποβάλει τα προγράμματα και να μας πείτε αυτά είναι κάντε ό,τι νομίζετε. Του είπα ότι θα ήταν σκόπιμο πριν ληφθεί η τελική απόφαση να υπάρχει τουλάχιστον μία άτυπη ενημέρωση. Του φάνηκε πολύ λογικό κατά πόσον θα το κάνει, δεν το γνωρίζω, ελπίζω να το κάνει γιατί αλλιώς στο τέλος του έτους θα υπάρξει εντονότατη αντιπαράθεση. Κάποιος είπε ο Χάνο ότι τα θέματα δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά θα τα καταφέρουμε να πείσουμε και εσένα, Χάνο. Ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και πάμε στον επόμενο Υπουργό που είναι αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Λοιπόν, τώρα ο Υπουργός Αθλητισμού και τουρισμού. Ο κύριος Φίσας έκανε την έκθεσή του για τον αθλητισμό σήμερα το πρωί μόλις. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα έχει πολύ χρήσιμα σχόλια. Αν είστε έτοιμος κύριε Υπουργέ, τότε έχετε και τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και χαρά η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Πολωνικής Προεδρίας για τον αθλητισμό. Μετά από τη σύντομη μου παρουσίαση, αν θέλετε, θα απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις, απορίες και σχόλια. Γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός για το Ευρωπαϊκό Κενοβούλιο και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι και η Πολωνική Προεδρία και εγώ ίδιος ατομικά και προσωπικά τη θέμεθα υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που οδήγησε σε μεγάλες προόδους στον αθλητισμό ιδιαίτερα μετά την εφαρμο... τη θέση ενισχύει της συνθήκης Λισαβόνας. Η Κομισιόν είχε κάνει τις πρώτες τις κατευθυντήριες γραμμές για τον συντονισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων και από τότε τον Μάιο το Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα εργασιών για τα επόμενα τρία χρόνια στον αθλητισμό. Η Πολωνική Προεδρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προτίθεται να εφαρμόσει αυτό το πρώτο πρόγραμμα εργασίας για τον αθλητισμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συγγράψει εκθέσεις που ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή από τον κύριο Σαντιάγο Πίσας και θα έχουν και αυτά τεράστια απήχηση. Εγώ έχω διαβάσει τις πρώτες εκδοχές του κειμένου και είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε ο αθλητισμός να γίνει μια σοβαρή και ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική. Η πολωνική προτεραιότητα στην Προεδρία της για τον αθλητισμό είναι το η εξής. Την, να αναπτυχθούν νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα του αθλητισμού μέσω της και αν εφαρμοστούν αυτές οι προτεραιότητες στους επόμενους 6 μήνες τότε η Πολωνία θα τονίσει ιδιαίτερα τα εξή θέματα. Πρώτον, η κίνδυνη που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός και η αθλητική πολιτική με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Γιατί τα διάλεξα αυτά. Γιατί η Ένωση πάνω απ' όλα πρέπει να υποστηρίζει τον αθλητισμό ως κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το είπαμε. Αλλά τα ιδεώδη του αθλητισμού και οι αξίες του θα ήταν ασήμαντα αν δεν υπήρχε ακαιρεότητα και τιμιότητα στον αθλητισμό. Γι' αυτό η Πολωνική Προεδρία θέλει να δώσει αγώνα για έναν καθαρό αγνό αθλητισμό. Θέλουμε να φανεί ότι ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός και για την οικονομία, διότι δεν δημιουργεί μόνο κόστος και δαπάνες αλλά και ωφέλη για τον υπολογισμό των κρατών μελών. Η στήριξη λοιπόν του αθλητισμού είναι και επένδυση. Το πρόγραμμα είναι πολύ φιλόδοξο. Και όπως είπα και πριν, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η κίνδυνη που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός. Μιλώντας για κινδύνους, εννοώ δύο πράγματα. Πρώτον, τα στημένα παιχνίδια και δεύτερον την, το τοπάρισμα. Αυτά είναι οι δύο μεγαλύτερες πληγές του αθλητισμού. Τα στημένα παιχνίδια σημαίνουν ότι ορισμένοι κερδίζουν κερδοσκοπικά. και επειδή τα τυχερά παιχνίδια και η κερδοσκοπία και η ηλεκτρονικά συνεχώς αυξάνονται, αυξάνονται και τα σκάνδαλα. Σκάνδαλα. Πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του αθλητισμού το ίδιο. Καταπολεμώντας τα στημένα παιχνίδια, Πρέπει να δούμε το πράγμα γενικότερα. Να απευθυνθούμε στις αθλητικές οργανώσεις και να θέσουμε και θέμα καλής διακυβέρνησης του αθλητισμού. Αυτό θα το πούμε στο, στη συνεδριάση του Συμβουλίου το Νοέμβριο. Νοέμβριο. Η Πολωνία θα προτείνει κατά τη συνεδρίαση εκείνη του Συμβουλίου τον Νοέμβριο καθώς προείπα do uznania oszustwa sportowego jako odrębnego przestępstwa kryminalnego w przepisach kraju. Όπως να θεωρηθεί το στημένο παιχνίδι ως εγκληματική παράνομη δραστηριότητα με να ζητηθεί ενισχυμένη συνεργασία με την αστυνομία και έρευνες για την διαφθορά αυτήν για να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα. Τα σώματα ασφαλείας και οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να συνεργαστούν μαζί με τις ε, οργανώσεις των στοιχημάτων. Νομίζουμε ότι θα είναι πολύ θετικό οι αρχές των χωρών μελών να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες που θα τους διατεθούν. διατεθούν. Ενώ παράλληλα θα διασφαλίσουμε το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων. E, Τέλος πάντων να καταπολεμήσουμε τις απάτες στον αθλητισμό και θα ζητήσουμε από τα καρά τη μέλη να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα πληροφόρησης, καμπάνιες πληροφόρησης για να γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι διαιτητές και οι διαιτήτριες, οι αθλητές και οι αθλήτριες, να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν αν σε περίπτωση που θεωρούν ότι κάποιο παιχνίδι είναι στημένο. Και θα συνεργαστούμε και με την Κομισιόν και τα οργανώσει των στοιχημάτων, ενώ υπολογίζουμε και στην υποστήριξη και στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερη απειλή κατά του αθλητισμού είναι το ντοπάρισμα. είναι και αυτό μια αθλητική απάτη διότι παραβιάζει το αθλητικό πνεύμα και καταστρέφει τα κίνητρα που μπορεί να είχαν οι τίμοι αθλητές και αθλήτριες. Καταστρέφει δε την εικόνα του αθλητισμού. Υπάρχουν εδώ και νομικά θέματα που τίθενται όπως η προστασία της ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων όπου χρειάζεται συντονισμένη αντιμετώπιση πανευρωπαϊκά για να καταπολεμηθεί το ντοπάρισμα στην Ένωση. Φυσικά θα συνεργαστούμε και με οργανώσεις αντιντοπαρίσματος για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει εκπροσώπηση της Ένωσης αυτές, να μιλούν όλοι με μία φωνή. Γι' αυτό η Πολωνική Προεδρία θα προετοιμάσει έναν δεοντολογικό κώδικα για το συντονισμό της ευρωπαϊκής θέσης για να για να συντονιστούν οι προσπάθειες από τη Διεθνή Οργάνωση Αντιντοπαρίσματος έτσι ώστε η Ένωση να εκπροσωπείται δεόντως. Άλλη προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας είναι η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι μια κοινωνική δραστηριότητα που βασίζεται πάνω απ' όλα σε εθελοντές και ερασιτέχνες βελτιώνει την κοινωνική ολοκλήρωση, συμπερίληψη και συνοχή. Και γι' αυτό η Πολωνική Προεδρία θα προετοιμάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το ρόλο του εθελοντισμού στον αθλητισμό και την προώθηση πιο ενεργού ρόλου των πολιτών. Το Νοέμβριο, το Νοέμβριο αυτά. Το έγγραφο εκείνο θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περισσότερο εθελοντισμό στον αθλητισμό και στοχεύουμε στη χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση αθλητικών γεγονότων στον τομέα του εθελοντισμού. Πράγμα που συμφωνεί και με το ότι φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Η Πολωνική Προεδρία είναι πεπισμένη ότι ο εθελοντισμός πρέπει να θεωρείται πολύ σημαντικός παράγων του αθλητισμού. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προτεραιότητα αυτή δεν περιορίζεται χρονικά γιατί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της ΟΕΦΑ το 12, θα βασιστεί στη δραστηριότητα εθελοντών και εθελοντριών και όταν λήξει αυτή η διοργάνωση θα πρέπει να δούμε τι πώς θα συνεχίσουν οι εθελοντές και εθελόντριες αυτές. Γιατί είναι εύκολο να τους βρούμε, αλλά μετά τι θα τους κάνουμε. Κατά την Προεδρία μας οργανώνουμε διάφορες διασκέψεις. Πρώτον, μία στις αρχές Ιουλίου για την ανατολική διάσταση της κινητικότητας Στις 18 και 19 Ιουλίου οργανώνουμε στο Βρότσουαλ μία διάσκεψη για τις ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό ως τμήμα της κοινωνικής πολιτικής πώς θα μπορούσε δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ιδιαίτερα ως προς αναπήρους, ε, ηλικιωμένους, μειονότητες γυναίκες. Τώρα για να επιστρέψω στον εθελοντισμό 13 και 14 Σεπτεμβρίου θα οργανωθεί στη Βαρσοβία διάσκεψη για τον εθελοντισμό στον αθλητισμό όπου θα μιλήσουμε για το ρόλο του εθελοντού ή της εθελοντρίας στις αθλητικές οργανώσεις και λέσχες. Ελάτε όλοι, σας καλούμε. Τέλος. Τελευταία προτεραιότητα, η αθλητική δραστηριότητα που βασίζεται σε οικονομικές πραγματικότητες. Καμιά φορά το ξεχνάμε ότι σε τέτοιες δύσκολες εποχές είναι και αυτό σημαντικό. Η Πολωνία αποφάσισε να τονίσει τη σημασία του αθλητισμού για την οικονομία. Θα τονίσουμε δηλαδή ότι αξίζει τον κόπο να στηρίξει κανείς τον αθλητισμό και οικονομικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι μόνο λόγω του πόσο σημαντικός είναι για την κοινωνία αλλά και για την οικονομία και για την παιδεία. Η Πολωνία λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει ένα δορυφορικό κανάλι όπου η Κύπρος, η Αυστρία δοκιμάσαν ένα τέτοιο κανάλι και τα αποτελέσματα ήταν θετικά και με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται ότι ο αθλητισμός δημιουργεί σχεδόν 2% του ΑΕΠ. Του ΑΕΠ. Θα σας δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία σε άτυπη υπουργική διάσκεψη στην Κρακοβία. Επίσης, υπάρχει τεράστια απήχηση του αθλητισμού οικονομικά και το αποτέλεσμα μιας σχετικής μελέτης θα για το πρωτάθλημα UEFA θα το πούμε επίσης στην Κρακοβία σε εκείνη τη διάσκεψη. Τώρα οι επιπτώσεις του αθλητισμού στην οικονομία είναι και θέμα χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει τον αθλητισμό να τον ε, συμπεριλάβουμε στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 14 με 20. Συμπεριλάβουμε. Ελπίζω η καλή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβουλίου να διασφαλίσει ότι και αυτή η πρόταση θα εφαρμοστεί απρόσκοπτα. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι το πρόγραμμά μας δεν πρόκειται να πετύχει παρά μόνο αν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη-μέλη και ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι αθλητικές οργανώσεις συμφωνήσουν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να ακούσω τυχόν σχόλια και απορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που παρουσιάστε με ε, Τέτοιο ενθουσιασμό τα θέματα του αθλητισμού. Εμείς ε, επιθυμούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα αθλητισμού. Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διαπιστώσαμε, τουλάχιστον ε, στο χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο μας έδειξαν, ότι εκεί αναφέρεται ο αθλητισμός Άρα δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάτι θα υπάρξει. Όλα αυτά όμως πρέπει να είναι σοβαρά γιατί όπως είπατε και εσείς ε, ο αθλητισμός ε, έχει πάρα πολλές ε, προεκτάσεις. Δεν είναι μόνο η αναψυχή των ανθρώπων. Έχει πολιτιστικές προεκτάσεις, προεκτάσεις στον τομέα της υγείας, πάρα πολλά θέματα. Η κυρία Μπόσκο. Κύριε Υπουργέ, ε, πρέπει να σας πω ότι με ικανοποιεί ιδιαίτερα το ότι εξηγήσατε με πολλές λεπτομέρειες ε, τις ε, προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία είπατε είναι πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τώρα τα στημένα παιχνίδια, το Νοέμβρη το Συμβούλιο θα αποφανθεί από αυτόν. Εγώ όμως θέλω να κάνω μία ερώτηση. Συμφωνώ ότι η απάτη στον αθλητικό χώρο είναι ποινικό αδίκημα, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να υπάρξει κάποια συμφωνία των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ε, αντιμετώπισης των ε, στημένων ε, παιχνιδιών. Σε κάποιες θεωρείται απάτη, σε άλλες ποινικό αδίκημα, σε άλλες παράπτωμα. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε κάποια λύση γιατί στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης διαχέονται αυτά τα σκάνδαλα. Τώρα είχαμε ένα στην Τουρκία αλλά και στη Φινλανδία και στην Ελβετία και εκεί υπάρχουν ε, προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το σημαντικότερο δυνατό. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, το Νοέμβρη θα είναι δυνατόν να γίνει μια βολιδοσκόπηση των κρατών μελών για να διαπιστωθεί ε, κατά πόσον ενδεχομένως ε, η Europol να επιληφθεί του θέματος. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει συνεργασία του οργανωμένου εγκλήματος, άρα δηλαδή πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει συντονισμένα τον, την αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να συνεργαστούμε με, τις ε, διάφορες, ε, με ε, φορείς που προσφέρουν τυχερά παιχνίδια. Οι περισσότεροι όμως βρισκόνται στην Ασία και είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε αυτούς. Σας ερωτώ λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτούς τους φορείς. Τρίτη ερώτηση, κώδικας κατά του ντόμπινγκ ντόπινγκ, αντιμετώπιση των αναβολικών. Ε, νομίζω ότι γίνεται λόγος για το θέμα ε, εδώ και πολύ καιρό. Ε, ορισμένα κρατημέλη πιστεύουν ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των πολιτών. Άλλοι πιστεύουν όχι, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση του ντόπινγκ. Εσείς τι πιστεύετε. Άλλη ερώτηση. Όσον αφορά τον αγώνα κατά του ρατσισμού, εμείς ε, πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού και ε, διακριτικής μεταχείρισης. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Σαντιάγο, ευχαριστώ πολύ, λέω και ο Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ καλές σας ιδέες για τον αθλητισμό. Ήδη συμφωνώ φάγαμε μαζί σας μια ομάδα ευρωβουλευτών με εσάς. Ε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρόσκληση. Όπως είπε η Πρόεδρος, αύριο θα παρουσιάσω την έκθεσή μου. Είναι μια έκθεση πιο περιορισμένη από ό,τι θα ήθελα, γιατί ε, το μέγεθος κάθε έκθεση είναι περιορισμένο. Ελπίζω με τις ε, ε, τροπολογίες θα συμπληρωθεί όμως. Χαίρομαι που λέτε, που είπατε ότι η Πολωνική Προεδρία ε, θέλει να προωθήσει την ποινικοποίηση της διαφθοράς στον αθλητισμό. Ε, όμως ε, ο ορισμός θα πρέπει να είναι ίδιος σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μόνον έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πρέπει να ορίσουμε πολύ καλά τι είναι αυτό το αδίκημα της διαφθοράς στον αθλητισμό. Επίσης μιλήσαμε για, την, ε, για τον αγώνα αντίον των αναβολικών, αντίον του ντοπαρίσματος. Αυτή η μάχη, αυτός ο αγώνας θα πρέπει να γίνει ε, με την... Ε, με το μέσο της καταπολέμησης των αναβολικών κάποιο άρθρο τη συνθήκη, το 80 τόσο, δεν θυμάμαι πιο ακριβώ είναι, μιλάει για τα φάρμακα. Θα μπορούσαμε εκεί, με βάση αυτό το άρθρο, να ε, αναλάβουμε δράση εναντίον των αναβολικών. Είπατε ότι το ντοπάρισμα είναι ε, απάτη, αλλά εκτός από απάτη είναι και αδίκημα κατά της υγείας. Και με ανησυχεί πολύ περισσότερο ε, το ντοπάρισμα ε, στα σχολεία, στα γυμναστήρια κλπ. και λιγότερο στα στάδια όπου υπάρχει και παρουσία γιατρών κλπ. Ε, θα πρέπει βέβαια όλος αυτός ο αγώνας να γίνει με σεβασμό στους αθλητές. Θα πρέπει να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά τους. Επίσης μιλήσατε, είπατε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ε, το βάρος που της ε, αξίζει στην Ουάντα και θα πρότεινα τη δημιουργία ενός ανώτερου δικαστηρίου, αθλητικού, ανώτερου δικαστικού, ανώτερου ε, αθλητικού δικαστηρίου στην Ευρώπη. Πώς ξέρετε υπάρχει ένα δικαστήριο στην Λοζάνη, σύμφωνα με την ελβετική δικαιοσύνη, που λειτουργεί σύμφωνα με την ελβετική δικαιοσύνη, η οποία βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ίδια με την κοινωτική δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα δικαστήριο τέτοιο τύπου δικαστήριο στις ΗΠΑ, ένα στην Αυστραλία, γιατί όχι και ένα στο Λουξεμβούργο. Επίσης, ε, κάνατε λόγο για την... Ε, ε, για τα δικαιώματα τις ε, διάφορες, ε, των διαφόρων ε, αθλητικών δραστηριοτήτων. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει σε πολλούς δημοσιογράφους, δεν αρέσει σε πολλά γραφεία στοιχημάτων, αλλά με την αναγνώριση αυτή της ιδιοκτησίας συγκεκριμένων αθλητικών εκδηλώσεων θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε και τον τοπάρισμα. Αυτό ε, μετά το άλλο θέμα που είναι ουσιαστικό είναι ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός και ο αεραστηχνικός αθλητισμός. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα σχολιάσω, δεν θέλω να μονοπολίσω το λόγο. Θα ήθελα απλώς να σας ρωτήσω ε, τι πιστεύετε για την υποστήριξη των αθλητών μας, η διπλή καριέρα, το έλεγα προηγουμένως και στην Υπουργό Άνωτερ της Εκπαίδευσης. Πολλοί από τους ε, αθλητές μας ε, θέλουν ε, όταν τελειώσουν την αθλητική τους δραστηριότητα να μπορούν να έχουν και ένα επάγγελμα. Επίσης να σας πω ότι με βάση τις, τις μελέτες που έχω εγώ διαβάσει ε, ο αθλητισμός αντιπροσωπεύει 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ε, το 3,65% του ΑΕΠ και το 5,4% του εργατικού δυναμικού. Όπως επίσης, επειδή είσαστε επίσης υπουργό τουρισμού, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη σχέση τουρισμού και αθλητισμού. Ε, τουρισμός και για την συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις και για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάκουλα παρακαλώ, σύντομα, να είστε σύντομος αν έχει την καλοσύνη. Εξ ονόματος εμού και της ε, δικής μου αθλητικής ομάδας των φιλελευθέρων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για αυτή την εξαιρετική παρέμβασή του. Καλύψατε όλους τους ε, τομεί που θα μπορούσε κανεί να φανταστεί, να σκεφτεί τους σχετικού με τον αθλητισμό. Και μια και δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, ο Σαντιάγο Φύσας ε, ετοιμάζει μια εξαιρετική έκθεση, ε, θα την ε, υποστηρίξουμε. Εγώ είμαι ταπεινός οπαδός σε αυτήν την περίπτωση θα ήθελα να επιμείνω όμως στο θέμα της διπλής καριέρας, τη δυνατότητα δηλαδή των νέων αθλητών να κάνουν και ε, να παρακολουθούν και σπουδές. Στα πανεπιστήμια και στι ανώτερε σχολέ ε, θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε την αθλητική ζωή όπως γίνεται στι ΗΠΑ με ε, ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, με εσωτερικούς αγώνες, αθλητικούς συλλόγους στα πανεπιστήμια κλπ. Ε, μιλήσατε για τις απειλές αλλά μιλήσατε και για τις ε, ε, ευκαιρίες του αθλητισμού και θα πρέπει να παρουσιάζουμε και την θετική ε, εικόνα του αθλητισμού, τα ωφέλη που έχει στην υγεία. Στο 99% των περιπτώσεων το αθλητισμός είναι θετικός, έχει ωφέλη για τον άνθρωπο. Μόνο το 1% είναι το, οι αρνητικές, οι σκοτεινές περιπτώσεις. Μετά μας μιλήσατε για όλα αυτά τα προγράμματα και επαναλαμβάνω μία ακόμα φορά το περιεχόμενο του προγράμματος είναι πιο σημαντικό από το όνομά του. Και μια και μιλάμε για τον αθλητισμό θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το Ειρήνα Σεβίνσκα ως όνομα ε, αλλά και του Άνταμ Μάλις, που είναι στην καρδιά όλων των Ευρωπαίων. Ε, τα προγράμματα, το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να είναι πραγματικά προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Άνταμ Μάλις, λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει όνομα για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Wir fliegen nur nicht zu hoch, sonst äh, kommen wir nirgends mehr an. Äh, Boris. O Boris έχει Dziękuję bardzo. Zgadzam się absolutnie z tą nazwą. Natomiast fakt... Κοιτάξτε, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε. Έχετε πάρει στα χέρια σας την έκθεση του συναδέλφου μας ε, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός για όλο τον τομέα. Γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός ε, χρειάζεται φιλόδοξους ε, στόχους και είναι απαραίτητο να υπάρξει ο συντονισμός που αναφέρεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταρτήσατε αυτό το τόσο φιλόδοξο σχέδιο. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε να είμαστε η φωνή του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Και επιθυμούμε ο αθλητισμός να προχωρήσει ως ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα ε, τα οποία παίζουν ε, νομίζω ρόλο σε σχέση με το πλαίσιο χρηματοδότησης. Νομίζω στην Πολωνία έλαβε πέρυσι η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 2.500 αθλητικές εγκαταστάσεις για παιδιά χρηματοδοτήθηκαν, αναγέρθηκαν και εκεί τα παιδιά μπορούν να αθλούνται. Βεβαίως ε, αυτό, αυτή η παρέμβαση πρέπει να γίνει και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω το εξής ε, στην, ε, στο πλαίσιο της πολιτικής ε, συνοχής. Έχουμε 400 δις για τις διάφορες περιοχές Ευρώπης. Εδώ λοιπόν ο αθλητισμός μπορεί να πάρει ένα κομμάτι. Ο αθλητισμός ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όλοι οι μαθητές στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε ε, καλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Και κάτι άλλο που ελέγχει. Έχουμε ένα ε, μεγάλο ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και αυτό θα μπορούσε να εκταμιεύσει χρήματα για αθλητές που βρίσκονται στο τέλος της αθλητικής, αθλητικής τους ε, σταδιοδρομίας. Οι αθλητές αυτοί με χρήματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να ακολουθήσουν μια άλλη καριέρα, να μετεκπαιδευτούν και νομίζω ότι εδώ εμείς μπορούμε να παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο και κατά τη διάρκεια της γιατί όχι. Βεβαίω, ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η έκθεση του Σαντιάγκο. Η συνάδελφο ε, Σενεσίν. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση του Υπουργού Γκρίς και τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για τον αθλητισμό. Αυτό που δεν καλύφθηκε είναι το εξής. Μιλήσαμε πολύ για την συμμετοχή, μιλάμε πολύ για τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Για παράδειγμα εισηγμένων εταιριών κλπ. Έχει αποδειχθεί ότι εκεί που υπάρχουν γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια, τα αποτελέσματα χρήσης είναι καλύτερα. Δυστυχώς στις, ε, στους αθλητικούς ομίλους δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Κάποιες ποσοστώσεις έχουν εισαχθεί, έχουν επιβληθεί, ε, αλλά η συνολική εικόνα δεν είναι θετική. Είμαι η συγκήτρια μιας νομοδότησης ε, που θα ληφθεί υπόψη από το Σαντιάγο, ε, εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών συγκεκριμένα. Και Σε αυτή τη γνωμοδότηση σχολιάζουμε το ποιο θα έπρεπε να είναι το ποσοστό των γυναικών ή η ποσόστοση των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια Αθλητικών Συλλόγων. Η ποσοτητα των γυναικων στα διοικητικα συμβουλια Προεδρία θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα καθόλου. Πόσο σας ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό. Γιατί τα γυναικεία ζητήματα δεν έχουν και πολύ μεγάλη παρουσία στις προτεραιότητες σας από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό για την παρέμβασή του. Ε, uh, δεν είναι εδώ το μόνο το πρόβλημα αυτό που έθεσε ο Υπουργός. Θέλω να ρωτήσω Ποιος είναι ο ρόλος του αθλητισμού, του μαζικού αθλητισμού, των μαζικών πρωταθλημάτων. Διότι υπάρχει το φαινόμενο της παχυσαρκίας στον πληθυσμό μας. Πώς βλέπετε λοιπόν το ρόλο των μαζικών, του μαζικού αθλητισμού σε σύνδεση και με τα σχολεία. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα, μια σύνδεση και με τον τουρισμό, ας πούμε ένας μαραθώνας στο Παρίσι, στη Ρώμη, στις Βρυξέλλες. Αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που κινούνται στην Ευρώπη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τη δημόσια υγεία και για το μέλλον της Ευρώπης γενικότερα. Σας κατευχαριστώ και σας εύχομαι καλή τύχη. Η κυρία Κώστα, σύντομα παρακαλώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η παρέμβαση του Υπουργού που εστίασε σε τρία θέματα. Τρία θέματα ουσιαστικά που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και την αθλητική πολιτική. Ε, συμφωνώ κυρίως αυτά που είπαν οι συνάδελφοι σε σχέση με τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης όπως είπε συνάδελφοι Φίσας, Κοσκούρτ και άλλοι. Περαιτέρω λοιπόν ενίσχυσης ε, της ε, δυνατότητας συνεργασίας, συντονισμού, ανταλλαγή απόψεων. Και αυτό που είπε επίσης ο κύριος Φίσας, ε, να υπάρχει εντός δικαστηρίου στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι αρμόδιο για παρανομίες στον αθλητισμό. Υπάρχει ας πούμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που μας δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό που είπατε και εντωμεταξύ σας μπορούν να υπάρξουν και κάποια ενδιάμεσα βήματα. Το δεύτερο που θέλω να πω η πρόσβαση στον αθλητισμό είναι ένα νέο δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Κατά την άποψη λοιπόν ερωτώ το εξής. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και κάποιους ε, δείκτες, δηλαδή πώς μπορεί ε, κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει μείωση της ε, εγκατάλειψης ε, του σχολείου. Αυτό έχουμε δείκτες. Πώς μπορούμε όμως ε, σε επίπεδο κρατών μελών να μετρήσουμε καλύτερα την συμμετοχή των πολιτών στον αθλητισμό. Να βρούμε κάποιους δείκτες όπως σας είπα. Γιατί από εκεί εξαρτώνται πάρα πολλά και για την υγεία και για πολλά άλλα θέματα συναφή με τον αθλητισμό. Κατόπιν είπατε ότι θα υπάρξει μια πρωτοβουλία εκ μέρου σα και ελπίζω να συμμετέχει και η δική μας Επιτροπή και άλλες επιτροπές πρωτοβουλία που θα αφορά στην ε, δυνατότητα ίσων ευκαιριών για όλους. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι κυρίως αναφορά το θέμα της αναπηρίας. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν ε, συγκεκριμένες συμβάσεις και ευρωπαϊκές ε, και των Ηνωμένων Εθνών που λένε ε, συμβάσεις που δυστυχώς δεν γίνονται απόλυτα σεβαστές. Υπάρχουν στοιχεία που τα αποδεικνύουν αυτό. Άρα και εκεί θέλω να τοποθετηθείτε. Να πω επίσης ότι όσον αφορά τον αθλητισμό θεωρώ ότι πράγματι και ο αθλητισμός πρέπει να ενταχθεί στη συνθήκη της Λισαβάνας. Όπως είπε η κυρία Πακ προηγουμένως, ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε κατά πόσον θα υπάρξει ουσιαστική χρηματοδότηση και ρωτώ, η Πολωνική Προεδρία θα ε, ασχοληθεί με το θέμα αυτό έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική επέμβαση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εάν γίνει κάτι τέτοιο θα ήθελα να είναι κάτι πέρα από αυτό που μπορεί να προσφερθεί μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για τις προτεραιότητές μας. Γιατί ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικό θέμα και για τη δική σας επιτροπή. Έχουμε όμως μόνο έξι μήνες, ενώ το πρόγραμμά μας είναι πολύ φιλόδοξο. Ελπίζουμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο να πετύχουμε στην επίτευξη των στόχων μας καθώς και των στόχων του κυρίου Φίσα. Οι προτεραιότητες μας συμπεριλαμβάνονται κατά κάποιον τρόπο και στην έκθεση του κυρίου Φίσα. Για τα στημένα παιχνίδια φυσικά είναι πρόβλημα διεθνές, όχι εθνικό και γι' αυτό η καταπολέμηση του είναι πιο δύσκολη από ότι καταπολέμηση του ντοπαρίσματος όπου είναι πρόβλημα πιο ατομικό. Τα στημένα παιχνίδια είναι τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος και επομένως απαιτείται συντονισμένη αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως και σε παγκόσμιο διαπλανητικό επίπεδο. Ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διασκέψεις, για συμβάσεις, κατά, για δημιουργία ιδρυμάτων αντι-doping. Υπάρχει ένα έγγραφο της Κομισιόν κατά του ντοπαρίσματος για συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Θα θέλαμε δηλαδή να υπάρξει ένας κοινό αποδεκτός ορισμός του τι είναι αθλητική απάτη. Η Πολωνία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και μερικές άλλες χώρες έχουν ήδη εγκρίνει κάτι τέτοιο ως ιδιαίτερη εγκληματική δραστηριότητα. Η Γαλλία και η Γερμανία το επεξεργάζονται ήδη και αυτό δείχνει ότι πολλά ευρωπαϊκά κράτη ήδη σκέφτονται μια τέτοια λύση. Θα θέλαμε και άλλα κράτη να ακολουθήσουν. άλλα. Τώρα για αυτά που είπε ο κύριος Φίσας, η έκθεση του όπως είπα και πριν συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους δικούς μας στόχους για την καταπολέμηση του ντοπαρίσματος πρέπει να θεωρείται σαν θέμα χρήσης ναρκωτικών και απαγορευμένων ουσιών γενικότερα. Η ιδέα αυτή ενός ευρωπαϊκού σε εισαγωγικά δικαστηρίου για το τοπάρισμα δεν είναι κακή ιδέα. Θα μπορούσε να λύσει πολλά προβλήματα μεταξύ των αθλητών και στη στηρίζουμε την ιδέα αυτήν. Για μας βέβαια ο εθελοντικός χαρακτήρας είναι το ουσιώδες. Η διπλή καριέρα των νεαρών αθλητών για την οποία μιλάμε ε, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Σε πολύ λίγες αθλητικές δραστηριότητες μπορεί ένας αθλητής να κερδίσει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να κερδίσει τη ζωή του μόνο από αυτήν. Ιδίως όταν λήξει η αθλητική του καριέρα. Πρέπει λοιπόν η λεγόμενη διπλή καριέρα να ενθαρρυνθεί. Αυτό το κάνουμε ήδη στην Πολωνία. Από την εκπαίδευση, από την παιδεία και φυσικά απαιτείται και συγχρηματοδότηση για την εκπαίδευση των αθλητών ώστε να βρουν κάποια δουλειά αφού λήξει η αθλητική τους καριέρα παραδείγματος χάρη στα πλαίσια του προγράμματος που αναφέραμε πριν και στο δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και μέσω της χρήσης του κοινωνικού ταμείου. Η αθλητική παιδεία κύριε Τακούλα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Είναι ο αθλητισμός πολύ σημαντικό θέμα για τους νέους στην κοινωνία μας. Εάν φανεί ότι κάποιος αθλητής ή αθλήτρια απεδείχθη απατεών, αυτό τα καταστρέφει όλα δεν υπάρχει πια αγνότης στον αθλητισμό. Η κυρία Σενίσιν μας μίλησε για τη συμμετοχή των γυναικών στα Συμβούλια Επιτήρηση Εποπτείας. Είναι δύσκολο εδώ να εφαρμόσουμε ποσοστώσεις. Εμείς θέλουμε γενικά καλή διακυβέρνηση και στα εθνικά και στα διεθνή σώματα. και πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση γυναικών γενικά σε αυτά τα σώματα. Γενικά. Έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετές και γυναίκες. Ο μαζικός αθλητισμός αναφέρθηκε από κάποιον ομιλητή εννοούσε μάλλον τον επαγγελματικό αθλητισμό εμείς υποστηρίζουμε πάνω απ' όλα τον αθλητισμό για όλους, για όλους και όλες. Δεν εννοούμε μόνο τον επαγγελματικό αθλητισμό, για όλους. Να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων, των παιδιών στα σχολεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια και ολόκληρες οικογένειες, ολόκληρες γενιές να συμμετέχουν, γονείς, παππούδες. Να είναι όλοι ενεργοί στον αθλητισμό τα μαζικά αθλητικά γεγονότα είναι κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Η κυρία Κώστα ρώτησε κάτι για την προσβασιμότητα να, είναι δήλα να διασφαλιστεί δηλαδή ο λαϊκός χαρακτήρας του αθλητισμού. Ναι, πρέπει να καταπολεμήσουμε τους φραγμούς δομικούς ιδίως. Πρέπει να υπάρχουν αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις δωρεάν για να είναι προσβάσιμες σε όλους. Ο κύριος Μπόρις μας είπε ότι στην Πολωνία οικοδομούνται στάδια και εγκαταστάσεις δωρεάν για όλους και όλες, ανοιχτά όλο το χρόνο. Και με τέτοια μέσα προσπαθούμε να αφαιρέσουμε, να περικόψουμε και οικονομικούς φραγμούς. Υπάρχει εδώ το πρόβλημα των αναπηριών και της ηλικία ορισμένων που θέλουν να αθληθούν αλλά το να είναι κανείς ε, αθλητής, το να αθλείται είναι κάτι που πολλές φορές απαιτεί και χρήματα. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την ύπαρξη τέτοιων οικονομικών φραγμών. Ελπίζω να απάντησα τώρα σε όλα αν όχι τα περισσότερα, σε περισσότερα αν όχι όλα τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε τις παρουσιάσεις της Πολωνικής Προεδρίας. Και είμαι βέβαιη ότι θα τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αντέξατε και θα τα πούμε σήμερα το απόγευμα ε, για την ακρόαση. Την ακρόαση δεν την κάνουμε για μένα, για, για όλους την κάνουμε, λέει η πρόεδρος. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι να έρθουν το απόγευμα. Και για αύριο το πρωί μην ξεχνάτε να φέρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ε, ε, θα σας το πω και απόγευμα, το απόγευμα. Να έρθετε λοιπόν το απόγευμα να το ξανακούσετε. Ευχαριστώ, καλή όρεξη, ευχαριστή τους ε, διερμηνείς πρόεδρος και οι διερμηνεί ευχαριστούν την πρόεδρο. Γεια σας.